Κυρίε και κύριοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε με μια μικρή καθυστέρηση, αλλά όσο το δυνατόν ε, γίνεται στην ώρα μας. Ε, και άμα σας ενοχλεί πείτε μου το, έτσι. Δεν είναι θέμα, θα σταματήσω. Αλλά κάποτε πρέπει να ξεκινήσουμε κιόλα. Έχουμε ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα, το γνωρίζετε. Ιτερ, Έχουμε υψηλού προσκεκλημένους, κάποιο λείπει ακόμα. Πρότασή μου είναι λοιπόν να ξεκινήσουμε τον Γενικό Διευθυντή της Διεθνής Έρευνας, τον κ. Σμίτς, σύντομα να μας ενημερώσετε πώς έχουν τα πράγματα. Δεν χρειάζεται τώρα ε, εξηγήσει για το πόσο σημαντικό είναι το ίτερ και τα λοιπά και τι δουλειά κάνει, τα ξέρουμε αυτά. Το θέμα είναι το πρόβλημα δηλαδή το ότι η Επιτροπή μας θέλει να συνεχίσει να υπάρχει το ίτερ και μετά θα αναζητήσουμε λύσεις για τα χρηματοδοτικά ε, ζητήματα. Αυτό πρέπει να λυθεί. Οπότε θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας βοηθήσει ως προς αυτό. Κύριε Σμίτς, λοιπόν, έχει τον λόγο. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είχα πει και την προηγούμενη επίσκεψή μου στην Επιτροπή σας ορίστηκα Γενικός Διευθυντής Έρευνα την 1η Ιουλίου. Η ΙΤΕΡ ήταν ο πρώτος φάκελος που έφτασε στο γραφείο μου και δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα που να μην τον βρω πάλι στο γραφείο μου. Θα σας κάνω κάποιες διευκρινήσεις σήμερα για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, ενώ οι συνάδελφοι ε, που ασχολούνται με τα δημοσιονομικά θα ασχοληθούν με αυτά. Εγώ θα ασχοληθώ περισσότερο με τη διαχείριση, την ε, καθοδήγηση και την ε, κατάσταση μετά την ολοκλήρωση για να δούμε και πώς θα, αποφύγουμε μελλοντικό κόστος. Οι κυβερνήσεις, ή μάλλον η δομή του ΙΤΡΕ είναι σύνθετη η... έχει την ευθύνη η οργάνωση Ήτρε για την δημιουργία και την επίδοση του μηχανήματος, ενώ τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν σε είδος τα διάφορα συστατικά μέσω των εθνικών εσωτερικών τους οργανισμών. Το Fusion for Energy είναι ο Ευρωπαϊκός Εσωτερικός Οργανισμός βρίσκεται στη Βαρκελόνα, Βαρκελόνη και βρίσκεται εδώ δεξιά, αριστερά μου ο Γενικός Διευθυντής του. Ε, προσφέρει πάνω από το 45% των πόρων στη φάρη της κατασκευής και, και 9% περίπου παρισσότερο από κάθε έναν από τους άλλους εμπλεκόμενους. Η Κομισιόν εκπροσωπεί την EU στο Συμβούλιο του ΣΥΤΡΕ που είναι το όργανο που διοικεί Ε, αλλά όλες οι αποφάσεις του οργανισμού απαιτούν ε, ομοφωνία. Αυτό συνεπάγεται μεγάλη εμπλοκή όλων των ε, συμμετεχόντων, αλλά και καλή οργάνωση και διοίκηση. Σε, τέτοιου βαθμού συνεργασία υπάρχει για κάποιος βαθμός περιπλοκότητας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το Fusion for Energy έχει υπάρξει μια, ως δημιουργηθεί ως κοινή επιχείρηση, η βασική της δραστηριότητα είναι να προμηθεύει και να προσφέρει στο ίτερ όλα τα στοιχεία του ίτερ που πρόκειται να παραδώσει η Ευρώπη. Πρέπει να εξασφαλίσουμε και αυτή τη στιγμή προβλέπουμε μέτρα για να ενισχυθεί η ε, δομή διοίκηση του έργου και σας έχουμε στείλει ένα έγγραφο εργασίας του προσωπικού που εγκρίθηκε πρόσφατα και που ξεκάθαρα προσδιορίζει πώς σκοπεύουμε να βελτιώσουμε την ε, δομή και την διοίκηση του έργου. Και βεβαίως ε, αναφέρομαι και στο διεθνές σκέλο, όσο και στο, στην κοινή επιχείρηση του Fusion for Energy που βρίσκεται στη Βαρκελόνη. Τώρα θα αναφερθώ στο ζήτημα του κόστους, που είναι και το δεύτερο θέμα που έχω στον κατάλογό μου. Όπως ξέρετε το έργο αυτό έχει αντιμετωπίσει σοβαρές αυξήσεις κόστους. Όμως πρέπει να σας θυμίσω ότι η ε, συμφωνία του υπογραφεί και το Νοέμβριο του 2006 επί τη βάση αρχικών εκτιμήσεων κόστους που έγιναν το 2001. Το 2001 και που στηρίχτηκαν από την ε, Επιστημονική Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Μία από τις πρώτες κινήσεις της ε, οργάνωσης ΙΤΡΕ που δημιουργήθηκε το 2007 ήταν ε, να πραγματοποιήσει μία σε βάθος λεπτομερή επανεξέταση του έργου που στηριζόταν, είπαμε το 2001, η οποία επανεξέταση οδήγησε στη σαφή διατύπωση ότι ε, χρειάζεται μία αναθεώρηση των, ε, του υπολογισμού του κόστους. Λόγω της, του μεγέθους της αύξησης του κόστους, η Κομισιόν αμέσως ζήτησε ανεξάρτητες εκτιμήσεις για, αυτές τις, ε, για αυτούς τους υπολογισμούς, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμους. Και μέχρι τα μέσα του 2009 όλες αυτές οι ανεξάρτητες εκτιμήσεις είχαν ολοκληρωθεί και γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά το ακριβές κόστος αυτού του ε, σε μεγάλο βαθμό διεθνούς έργου, τα οποία βεβαίως αμέσως ε, σας γνωστοποίησαμε. Χάρη στην τεράστια αύξηση του αυτού του κόστους, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ένα χάσμα χρηματοδότησης για το ΙΤΡΕ, 1,4 δις. Και κάνουμε μια πρόταση πώς να βρεθούν αυτά τα κεφάλαια που λείπουν. Θα ακούσετε περαιτέρω από τους συναδέλφους. Όσον αφορά την διοίκηση του έργου αυτού, η Κομισιόν προτείνει τρόπους και δραστηριότητες για να εξασφαλίσουμε μια ισχυρότερη διοίκηση. Είναι μια σημαντική πρόταση της Κομισιόν που υποστήριξε και όχι μόνο αφορά αυτό την λειτουργία του οργανισμού Fusion for Energy αλλά και τον διεθνή οργανισμό μας είπαν ότι έχει αντικατασταθεί και στους δύο οργανισμούς η ανώτατη διοίκηση. Και τώρα έχουμε δύο πρώτης τάξεως ε, managers οι οποίοι έχουν αποδείξει τις διοικητικές τους ικανότητες σε διεθνές επίπεδο. Ο Φρανκ Βρίσκο στη Βαρκελόνη, Fusion for Energy, και ο καθηγητής μου το Χήμα, γενικός διευθυντής του Ήτρε στο Κανταχάσου ο κύριος Μπρίσκο κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσει ο οργανισμός Fusion for Energy να ανταποκριθεί στους σκοπούς του. Να γίνει δηλαδή ο οργανισμός αυτός λιτός, αποδοτικός, αποτελεσματικός, να εξυπηρετεί το σκοπό του για να μπορέσει να αναλάβει, να διοικήσει αυτό το τεράστιο έργο. Το έγγραφο εργασία του προσωπικού που σα στείλαμε χθε το βράδυ εξηγούμε λεπτομερώς τα διάφορα μέτρα που σκοπεύουμε να πάρουμε για να δείξουμε ότι μόνο ένα είναι ο σκοπός μας, δηλαδή να αποφύγουμε ε, την, την υπερβολικό κόστος στο μέλλον και να υπάρχει μια καλή διαχείριση αυτού του έργου, καλή διακυβέρνηση, πράγμα που χρειάζεται οπωσδήποτε για να αντιμετωπίσουμε ε, τους φιλόδοξους στόχους μας στον τομέα της ενέργειας και των, της μείωσης του διοξιδίου του άνθρακα. Ο Φρανκ Μπρίσκο βρίσκεται εδώ δίπλα μου, ήδη έχει προετοιμάσει ένα φιλόδοξο ε, πρόγραμμα δράσης. Ήδη είδαμε κάποια από τα αποτελέσματά του Ήδη ε, είδαμε τα πρώτα μέτρα που βελτιώνουν τις διαδικασίες κρατικών προμηθειών, περιορίζουν το κόστος και αργότερα θα, θα έχει τη δυνατότητα, ελπίζω κύριε Πρόεδρε, να πάρει και αυτό το λόγο για να σας δείξει ότι πράγματι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να βελτιωθεί η διοίκηση αυτού του σύνθετου διεθνούς έργου. Σας ευχαριστώ. Mit Blick auf die Uhr möchte ich als nächsten Herrn Generaldirektor für den Haushalt, Herr ε, Βλέπουμε λοιπόν ε, το Γενικό Διευθυντή για τον Προπολογισμό, τον κύριο Ζανζάν, τον, στον οποίο θα ήθελα να δώσω τον λόγο γιατί θα πρέπει και μισή να φύγει για άλλη διαπραγμάτευση. Οπότε έχετε τον λόγο κύριε Ζανζάν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα της ε, χρηματοδότησης ε, ε, αυτού του 1,4 δις επιπλέον δαπάνης από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπαθήσαμε να ταυτοποιήσουμε σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο δημοσιονομικό περιβάλλον τα μέσα εξέβρεσης κατάλληλης χρηματοδότησης ώστε να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη αυτή. Παρουσιάσαμε τον προηγούμενο Ιούλιο μια ανακοίνωση προς το Συμβούλιο που θα πρέπει να τοποθετηθεί στη συζήτηση με τα κράτη-μέλη ε, εν ώψη της ε, προεδρίας, ε, συγγνώμη, εν της προετοιμασίας που κάναμε για τον προηγούμενο Ιούλιο, καθώς και στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, μια πρόταση χρηματοδότησης για τα έτη 2012-2013, χρηματοδότησης λέω, των, των ε, ε, αναγκών, των κονδυλίων ε, υποχρεώσεων από 860 εκατομμύρια ευρώ, γνωρίζοντας ότι δεν έχουμε ακόμα βρει την χρηματοδότηση για 540 εκατομμύρια. Τα 860 εκατομμύρια για τα οποία ήδη κάνουμε συγκεκριμένη πρόταση, σε αυτά 400 εκατομμύρια προέρχοντο από το διαθέσιμο, ε, προ, ε, από το διαθέσιμο της γραμμής 2 ε, και 460 που προέρχοντο από την αναμόχλευση του κεφαλαίου Α που αφορούσε αύξηση των δεσμεύσεων κατά ένα δις ευρώ. Έκτοτε κάναμε μια νέα εκτίμηση των αναγκών μας, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη το αίτημα, το πιεστικό από το Συμβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να δώσουμε συγκεκριμένη περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ε, προτιθέμεθα να δώσουμε την ολοκληρωμένη χρηματοδότηση. Η κατάσταση, κυρίως ε, όσον αφορά το κεφάλαιο 2, μας ε, επιτρέπει το ενδεχόμενο ουσιαστικής επιπλέον χρηματοδότησης πάντα με, από το κεφάλαιο 2 μέσα από μεταφορά ε, διαθέσιμου αποθεματικού. Προς το 1α και εν συνόλο Εάν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο το δεχτούν, μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ήδη στα πλαίσια της δημοσιονομικής ε, διαδικασίας, της ισχύουσας διαδικασίας ε, και όσον αφορά και τον διορθωτικό προϋπολογισμό του 2010, ε, το είναι η χρηματοδότηση του 1,4 δις με κατανομή ως εξής, μεταφορά από το 2 ύψους 814 ε, εκατομμυρίων ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τα, τις ε, διαθέσιμες, τα τους διαθέσιμους πόρους μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού, 93 εκατομμύρια από το κεφάλαιο 5, διοικητικές δαπάνες και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη τις ε, αξιολογήσεις ε, μισθολογικής ε, προσαρμογής που θα μειωθούν όσο γίνεται περισσότερο. Υπάρχουν προοπτικές εξοικονόμησης της τάξεως των 54 και 39 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή εξοικονόμηση 93 εκατομμύρια το μισολογικό κόστος. Έχουμε επίσης 18 εκατομμύρια στο 4 και 15 εκατομμύρια στα πλαίσια του 1α με αναμόχλευση έτσι όπως την έχουμε προβλέψει. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε συνολικά να απαντήσουμε στην ανάγκη χρηματοδότησης για το ίτερ ήδη από το φθινόπωρο. και επομένως ε, να είμαστε σε θέση να δώσουμε συνολική απάντηση και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω τίποτα άλλο, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Είναι σημαντικό το σύνολο των διατάξεων αυτών να εγκριθεί άμεσα, ήδη από τώρα, γιατί έχουμε το διορθωτικό προπολογισμό του 2010 και το προσχέδιο του προπολογισμού του 2011. Τα πράγματα αλλάζουν διαρκώς ε, και αν ε, περιμένουμε να χρηματοδοτήσουμε το ίτερ ε, από τα μέσα τα οποία τώρα ε, ε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε θα αντιμετωπίσουμε τελικά μεγάλο πρόβλημα γιατί δεν θα υπάρχουν διαθέσιμα ε, κεφάλαια στον προϋπολογισμό του 2011 και αυτό θα είναι μεγάλο πρόβλημα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τέλος θα ακούσουμε τον Διευθυντή της Υπηρεσίας στη Βαρκελόνη, τον κύριο Μπρίσκο για μια σύντομη τοποθέτηση. Σύντομα για να κάνουν και ερωτήσεις συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλη χαρά θα κάνω μια μικρή εισαγωγή. Κυρίως για δύο πράγματα θα μιλήσω. Οι επόμενες μέρες της δραστηριότητας του Ήτρε και η πρόοδος που θα γίνει. Είναι μια τεράστια επιστημονική επιχείρηση, όμως τα επόμενα ε, νέα δέκα χρόνια είναι ένα κατασκευαστικό έργο. Πριν φτάσω στη Βαρκελόνη ήμουν είχε γίνει μια εξωτερική αξιολόγηση που έλεγε ότι δεν υπήρχε αρκετή τεχνογνωσία στον τομέα του project management στη Μαρκελόνη και συμφώνησα απόλυτα και έκανα προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο που εγκρίθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου για να, ώστε να αλλάξουμε τα πράγματα, πράγμα που ήδη έχει ξεκινήσει. Οπότε, άλλαξα τη δομή, πρόκειται, έχει τώρα... Ε, ε, γίνει, έχει αποκτήσει τη μορφή ομάδων έργου που έχει ε, συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Άλλαξα κάποιες από τις διαδικασίες του project management και εισήγαγα και κάποιες ε, βιομηχανικές διαδικασίες και πριν το τέλος του μήνα οι επικεφαλής αυτών των ομάδων έργου θα συναντηθούμε για να εξετάσουμε το, την κατάσταση και τέλος μετά από αυτό ίσως χρειαστεί να αλλάξει ένα μέρος του προσωπικού. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι των ομάδων ε, των έργων αυτή τη στιγμή ε, εκτελούν υπηρεσιακά χρέη και μπορεί να προσληφθούν άλλοι. Ένα άλλο θέμα που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι το ΙΤΕΡ προχωρεί αυτή τη στιγμή ξεκίνησε με βραδείς ρυθμούς το 2007. Όλοι δυστυχώς ε, υποτιμήσαμε πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να συσταθεί ένας τελείως νέος οργανισμός τόσο στο Κάβερας και όσο και στην Βαλκελόνη και έλειπε και ο σχεδιασμός, ε, δεν είχε απολύτως ολοκληρωθεί. Το διάστημα αυτό πλέον ολοκληρώθηκε, πέρασε και φέτος περάσαμε στην πραγματική κατασκευαστική φάση. Έχουμε ήδη ξεκινήσει, ε, συνάψει βασικά, βασικές συμβάσεις για βασικά ε, στοιχεία του, του έργου. Μέχρι το τέλος του 2010 θα έχουμε ε, συνάψει συμβάσεις για περίπου 20 δις δολάρια που, εξωτερικής, εξωτερικών ε, δουλειών, ε, δουλειάς που θα είναι περίπου το 25% του συνόλου της αν πάτε στο Κανταράς θα δείτε ότι η κατασκευή έχει ήδη ξεκινήσει, οι σκελετοί κάποιων μεγάλων κτηρίων ήδη υπάρχουν και η δουλειά προχωρεί με καλούς ρυθμούς. Εκ παραλίλου ξεκινήσαμε τις, ε, τις συμβάσεις με διάφορα ε, διάφορες μονάδες στην Ευρώπη για τα βασικά στοιχεία, τους μαγνήτες δηλαδή και την φάση του κενού. Δηλαδή ήδη έχουμε περάσει την κατασκευή, αυτό θέλω να σας διαβεβαιώσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα θα ακούσουμε βεβαίως τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, τον κύριο Λαμό. Ίσως θα θέλατε να πείτε λίγα λόγια. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κύριε Γενική Διευθυντά, κύριε Διευθυντά, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που προσκαλέσατε την Προεδρία στη συζήτηση αυτή. Θα είμαι πολύ σύντομο. Όπως γνωρίζετε, στις 12 Ιουλίου το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα στα οποία ξεκάθαρα διατύπωσε τη σημασία της πρόοδου του έργου ΙΤΕΡ. Αυτό όμως συνεναρτάται με διάφορες προϋποθέσεις, δηλαδή επιπλέον ε, ανάγκες στην περίοδο 2012-2013 και γι' αυτό το Συμβούλιο προτίμησε την τήρηση του υφιστάμενου ορίου του πολιετούς προγραμματισμού από το 1α, λαμβάνοντας υπόψη πρώτον τα μη ε, χρησιμοποιηθέντα κονδύλια και δεύτερον ε, επιβάλλοντας μια καταποκοπήν βάση και κάνοντας τους απαραίτητους προσαρμογέ. Ε, τις απαραίτητες προσαρμογές και βεβαίως τα ποσά θα καθοριστούν στη βάση των ε, ε, δημοσιονομικών συζητήσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει. Χθες για πρώτη φορά συζητήσαμε την, ε, στον τριμερή διάλογο την χρηματοδότηση του ΙΤΕΡ. Υπάρχουν κάποια στοιχεία αριθμητικά η Προεδρία σας διασφαλίζει ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε την ταχύτερη δυνατή πρόοδο. Η Προεδρία ε, συνεργάζεται με την Κομισιόν που, παίζει το, διευκολύνει αυτές τις συζητήσεις. Ως Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου για την έρευνα και τα θέματα ατομικής ενέργειας θα σας διαβεβαιώσω ότι το ε, σχέδιο ελέγχου του, των αποφάσεων, το σχέδιο αυτό θα εγκριθεί από το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα και έρευνα στι 26 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει την δική τη πρόταση μεταρρύθμιση για την διακυβέρνηση του ε, έργου ΙΤΕΡ. Σα ευχαριστώ για την προσοχή. Ähm, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα θεσμικά όργανα εδώ πέρα δηλώνουν πως ε, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον ε, για να συνεχίσει να λειτουργεί και να εξελίσσεται το ίτερ αλλά επίσης δηλώνουν πως ε, είναι και προς το συμφέρον μας να γίνει αυτό με τρόπο οργανωμένο. Ε, πέντε συνάδελφοι μου ζητήσαν λόγο. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να προσπαθήσετε να είστε λίγο σύντομοι γιατί ο κύριος Ζανζόν πρέπει να πάει και κάπου αλλού. Αν υπάρχουν λοιπόν ερωτήσεις που απευθύνονται απευθείας προς τον κύριο Ζανζόν, σας παρακαλώ να μας το πείτε για να ακουστούν αυτές πρώτες. Αλλιώς θα πάρετε το λόγο με τη σειρά που αναφέρετε εδώ πέρα. Η Ριέρα Μαδουρέλ πρώτα απ' όλα. Δέκα έγιναν το μεταξύ συνάδελφοι. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίζω τους τέσσερις ε, προσκεκλημένους μας ε, και τους ευχαριστώ. Όπως είπε ο πρώτος, πράγματι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο αυτό, το οποίο μόλις τώρα βεβαίω, ε, με το οποίο μόλις τώρα εξοικειωθήκαμε και το στηρίζουμε, αλλά έχουμε διάφορα προβλήματα, οικονομικά, προϋπολογισμού, διαχείρισης, πάρα πολλά όπως μας είπατε. Και Ακόμα και όσοι είναι υπέρ του προγράμματος ανησυχούν. Τώρα ξέρουμε τα προβλήματα, πρέπει να δούμε ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν στο οργανόγραμμα και στις διάφορες αρμοδιότητες. Το ερώτημα μου κύριε Σμίτ είναι για να υπερασπιστούμε αυτό το μοντέλο. Τι έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο, του τελευταίους μήνες για να διασφαλίσουμε πως το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να σας εμπιστευτεί ξανά. Τι θεωρείτε πως έχει γίνει σωστά μέχρι τώρα και τι θα γίνει σωστά στο μέλλον. Βεβαίω. Πρέπει να δούμε και τα νούμερα, δεν μπορώ να πω τίποτα αυτή τη στιγμή για τον προπολογισμό, αλλά πρέπει να ξέρω τι θα κάνετε στο μέλλον για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη. Κάτι άλλο μας φάνηκε περίεργο, δεδομένου του ότι είναι ένα τόσο σημαντικό έργο και έχει τόσο μεγάλη οικονομική σημασία και έχουμε τόσα προβλήματα με τη νέα οργανωτική δομή, με τη Γιουρατόμα και με τον νέο Γενικό Διευθυντή. Πού βρίσκεται το έργο στο πλαίσιο της γιουρατόμ, Κρίστιαν Χέλλερ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Πρώτα απ' όλα, να πω το εξής, ναι, η πλειοψηφία των βουλευτών υποστηρίζουν το ίτερ. Πρέπει όμως να πω πως αυτό δεν είναι ανεφόρον. Τρεις πτυχές είναι σημαντικές. Πριν από δύο ώρες λάβαμε το έγγραφο στο οποίο η Κομισιόν μας παρουσιάζει και τις μελλοντικές της ιδέες για την διαχειριστική δομή στο διεθνές επίπεδο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στο επίπεδο της σύνδεξης για την ενέργεια, το, του Fusion for Energy. Υπάρχουν κάποιες πτυχές για την ευρωπαϊκή διαχείριση, ε, τις οποίες αναφέραμε σε ένα υπερκομματικό νομίζω έγγραφο και λέμε πως πάμε προς σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να πούμε πως όλα αυτά είναι σχέδια μέχρι στιγμής, γιατί άκουσα τους εκπροσώπους της διοίκησης που λένε πως ε, τώρα ξεκινήσαμε. Δεν έχετε ξεκινήσει. Και εδώ πέρα έχει τη σημασία του προπολογισμού. Δεν νομίζω πως το κοινοβούλιο χωρίς να ξέρει ποιες είναι οι νέες δομές, ποιος είναι ο μηχανισμός ελέγχου, μπορεί να κάνει να δώσει μια υπόσχεση όσον αφορά τον προπολογισμό. Δεν είναι δύο ξεχωριστέ διαδικασίες, γιατί ε, αυτές οι διαδικασίες είναι υπό αυτή την αίρεση. Να δώσω ένα παράδειγμα γιατί ακούστηκε πως ε, τα νούμερα είναι του 2001 και βεβαίως τώρα θα είχαμε διαφορετικά νούμερα. Αυτό δεν το αμφισβητήσαμε ποτέ. Απλά διαβάσαμε και τα δικά σας τα πρακτικά και ο έλεγχος απέτυχε ακριβώς γιατί έπρεπε να γνωρίζετε ήδη σε αιτήσια βάση την απόκληση. Το ότι γίνεται πιο ακριβό το έργο είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό, αν και δύσκολο από πλευράς του υπολογισμού, αλλά γιατί επί σειρά ετών ε, δεν είχατε κάποιον έλεγχο για την απόκληση αυτή, είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε και αυτό είναι και θέμα του δικού σας εσωτερικού ελέγχου, τον οποίο διαβάσαμε, τον οποίο είχε η διοίκηση εδώ και καιρό και η Κομισιόν εδώ πέρα ε, δεν είδε τα λάθη στον έλεγχο και κάποιες περιπτώσεις οι οποίες είναι αμφίβολες θα πω. Στον προπολογισμό έχουμε ένα βασικό πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα είναι σωστά τα νούμερα γιατί τα νούμερα βασίζονται στο ότι δήλωσε το Συμβούλιο τον Ιούλιο ότι δεν θα δώσει 7,2 δισεκατομμύρια αλλά 6,6. Αυτά είναι ευσεβείς πόθη και είπε το ΔΣ πως τα καταφέρνουμε και με 6,6 δισεκατομμύρια. Γιατί γίνεται αυτό, κανείς δεν μας είπε ποιο είναι το περιθώριο λιγμών που υπάρχει για χρηματοδότηση σε αυτό το επίπεδο. Δεύτερον, όσον αφορά τον άμεσο προϋπολογισμό, Τώρα μας λένε πως ε, στο τέλος Νοεμβρίου πρέπει να δώσουμε τα λεφτά γρήγορα γιατί του χρόνου δεν θα υπάρχουν. Να σου το πω σαφώς, δεν θεωρώ πως είναι διατεθειμένο να το δεχτεί αυτό το κοινοβούλιο χωρίς να οριστεί ποιες είναι οι νέες δομές. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε μεταφορές ε, στον προπολογισμό από τον πυλώνα 1α που είναι το 7ο ε, πρόγραμμα έρευνα ή ευρατόμα αντικείμενο διαπραγμάτευση δηλαδή του προπολογισμού χωρί να ξέρουν ποιε είναι οι νέε διοικητικέ δομέ και αν είναι σωστά τα νούμερα. Δεύτερο πρόβλημα. Δεν έχουμε μόνο το θέμα της υποχρηματοδότησης τα επόμενα δύο χρόνια, αλλά η διεθνή δομή είναι έτσι ώστε κατά βάση δεν ε, ορίζει ο Διεθνής Οργανισμός τα τεχνικά στοιχεία, αλλά οι εθνικές υπηρεσίες. Και το έχουν πει αυτό και οι εμπειρογνώμονες πως ε, αυτό θα οδηγήσει σε επιπλέον κόστος εκτός αν αλλάξει η διεθνής αυτή διακυβέρνηση. Οπότε το ερώτημα είναι πώς θα πρέπει να χρηματοδοτούμε στο μέλλον Δηλαδή πάλι αυτό το επιπλέον κόστος θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα πλαίσιο 7 ή 8 ή 18 ή θα έπρεπε η Κομισιόν να δει πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτή την αύξηση του κόστος και όχι μόνο για το ITER αλλά και για το Γαλιλαίο και το GMES για να τα εξορροπήσουμε αυτά στον προπολογισμό γιατί μπορεί ίσως αυτή τη στιγμή να χρηματοδοτήσουμε αυτό το έλλειμμα για δύο χρόνια από τα λοιπά του τίτλου 2, αλλά δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό στο μέλλον χωρίς μεγάλες περικοπές στο ερευνητικό πρόγραμμα. Οπότε τα ερωτήματα τα τρία είναι πρώτον, υπόσχεση για τον προπολογισμό μπορούμε να τη δώσουμε μόνο με δέσμευση για το ποια θα είναι η μελλοντική δομή τη διοίκηση και μη μου λέτε πώ την έχετε ήδη εφαρμόσει γιατί δεν ισχύει. Δεύτερον, τι θα κάνουμε με τα προβλήματα τα οποία δεν είναι ευρωπαϊκά αλλά θα προκύψουν στο μέλλον από το διεθνές επίπεδο που ξέρουμε πώς θα προκύψει επιπλέον κόστος. Πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά στον προπολογισμό και τρίτον, πρέπει να το πω αυτό, χρειαζόμαστε να μας πείτε πώς εντάσσονται αυτά τα μεγάλα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου 7. Ε, γιατί εντάξει μπορεί να βρούμε τα λεφτά για το ίτερ αλλά δεν ξέρουμε που θα βρούμε για τα άλλα έργα. Και αυτά είναι τα ερωτήματα που σχετίζονται με το ίτερ. Ευχαριστώ και όταν Σίσελη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να πω κάτι αντίστοιχο με τον προαναλύσαντα συνάδελφο και θα είμαι και πάρα πολύ σύμφωνη. Συμφωνώ το σχέδιο, το πρόγραμμα πρέπει να προχωρήσει. Δεν μπορεί να πούμε όμως ε, ότι... Ε, λείπουν τέσσερα δις και κάπου πρέπει να τα βρούμε. Πρέπει να συζητήσουμε για τις προϋποθέσεις ε, βάσει των οποίων θα εγγυηθούμε τα τέσσερα δις αυτά. Θα ήθελα να έχω από την Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με το πώς θα εγγυηθεί αυτές τις ε, προϋποθέσεις και τους ε, όρους. Ας πούμε, ο νέος υπολογισμός των τιμών θα πρέπει να είναι ακριβής έτσι ώστε ε, να δημιουργηθεί και ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Επίσης, καλό θα ήταν να λύσουμε όσο γίνεται περισσότερα προβλήματα ήδη από τώρα. Ε, όσον αφορά τώρα το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, έχουμε κάποιες επιφυλάξεις και ο υπολογισμός θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να μην υπάρξουν υπερτιμολογήσεις αργότερα. Χρειαζόμαστε ε, σαφές πρόγραμμα, σαφές χρονοδιάγραμμα και μια καλά καθορισμένη διοικητική δομή έτσι ώστε ε, όλα να γίνουν με σαφήνεια και ακρίβεια χρονική. Ενδεχομένως οι λύσεις και οι απαντήσεις να βρίσκονται στο έγγραφο το οποίο ε, αναφερθήκατε εσείς, αλλά δυστυχώς εγώ δεν μπόρεσα να μελετήσω το έγγραφο αυτό, δεν το είδα καν, ίσως να έφτασε ε, λίγο πριν ε, τη συζήτησή μας, αλλά κοιτάξτε, αυτό δεν είναι και τόσο σοβαρό. Πολύ καλύτερη θα ήταν η κατάσταση εάν είχαμε την δυνατότητα πρώτα να διαβάσουμε το έγγραφο και μετά να διατυπώσουμε ερωτήματα. Δεύτερο μιλήσατε, αναφερθήκατε στην, ε, αναφερθήκατε λέω στην αλλαγή διοίκησης ε, στο Fusion for Energy. Πώς μπορεί να έχει εμπιστοσύνη η Κομισιόν ε, στην δομή αυτή και στο μέλλον. Ευχαριστώ η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αυτό το πρόγραμμα ITER είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο είμαστε και εμείς εταίροι. Και επομένως ως εταίροι δεν μπορούμε παρά να στηρίξουμε πλήρως και ουσιαστικά ένα τέτοιο σχέδιο το οποίο ε, αναφέρεται στο μέλλον γιατί βεβαίως οι μελλοντικέ γενιές είναι αυτές οι οποίες θα ωφεληθούν από αυτό το ε, ε, πρόγραμμα. Αλλά θα πρέπει όντω ω πολιτικοί να μην βλέπουμε μονάχα το σήμερα ή το αύριο, αλλά και να έχουμε πιο μακρόθωρη προοπτική. Το κόστος ε, που ανακοίνωσε το ίτερ είναι μεγάλο. Μας έδωσε η Επιτροπή κάποια ε, στοιχεία και ανακουφίζομαι λίγο βλέποντας ότι υπάρχουν κάποιες λύσεις στον προϋπολογισμό 2010 έτσι ώστε να δοθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα μπορούσαμε να πούμε δεν συμφωνούμε, δεν ε, συμφωνούμε, δεν δίνουμε την σύμφωνη γνώμη μας για το επιπλέον πόσο αυτό θα σήμαινε ότι δεν θέλουμε θέλουμε να συνεχίσουμε να παίζουμε με τους εταίρους μας. Και τότε οι εταίροι μας πώς θα μπορούσαν να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι εδώ ε, πρόκειται για ένα ζήτημα αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλο τον κόσμο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια, να φύγουμε από αυτή την αχλή οποία, η οποία μας δυσκολεύει όλους. Οπωσδήποτε σε αυτό το πρόγραμμα ITER δεν υπήρξε η διαφάνεια, δεν υπήρξε η απαραίτητη επικοινωνία. Καταλαβαίνουμε βεβαίως ε, τις δεσμεύσεις του προϋπολογισμού. Βεβαίως τα στοιχεία τα οικονομικά του 2001 δεν μπορεί να είναι ίδια με το 2010 ή το 2011. Ε, υπάρχουν αυξήσεις οι οποίες ε, είναι απολύτως εξηγήσιμες, αλλά θα έπρεπε να είχαν εξηγηθεί αυτά τα επιπλέον κόστη σιγά σιγά στη διάρκεια των ετών, έτσι ώστε ο όλοι να ξέρουν στο τέλος ε, τι τους περιμένει. Και βεβαίως ε, όταν έγκαιρα ε, λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις, έγκαιρα μπορούν να προγραμματιστούν και κάποιες ε, κάποιες ε, ε, αποταμιεύσεις, κάποιες εξοικονομήσεις μάλλον. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι δυνατόν να ουσοδρομήσουμε όσον αφορά ένα τέτοιο πρόγραμμα. Πρέπει να συνεχίσουμε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει. Αλλά για να γίνει αυτό, για να συνεχίσουμε λοιπόν με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει, χρειαζόμαστε πλήρη διαφάνεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας εξήγησε ότι έχει λύση έτσι ώστε να εξευρεθούν τα απαραίτητα κονδύλια. Το καταλάβαμε αυτό, αλλά βεβαίως θα πρέπει να βιαστούμε, να αποδεχτούμε τις προτάσεις αυτές. Και εγώ θα ήθελα να μην είναι ε, μονάχα ε, να περνάει από το χέρι μόνο της Επιτροπής Προϋπολογισμών το εάν θα περάσει αυτό το σχέδιο ή όχι. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ε, η έρευνα είναι μακροπρόθεσμη επένδυση και ειδικά από αυτό θα ωφεληθούν τα εγγόνια μας, ούτε καν τα παιδιά μας. Είναι ένα ρίσκο που πρέπει να διατρέξουμε. Πράγματι αυτό το οποίο υπόθηκε για το καταράσμα γιατί πήγα εγώ, ε, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και νομίζω πως αποτελεί ένα ορόσημο και υποδειγματικό έργο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Πρέπει να πάμε όλοι και να δούμε γιατί μιλάμε. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε πώς πράγματι είναι ένα έργο στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πρωτοποριακό ρόλο και δεν πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό. Ο Ζανζόν παρουσίασε το κ. Ζανζόν τις ιδέες του και πράγματι θα πρέπει να αναλάβουμε τα βήματα εκείνα τα οποία πρέπει. Υπάρχουν τρόποι χρηματοδότησης. Επίσης πρέπει να πούμε πως η δημοσιονομική πειθαρχία δεν ήταν η καλύτερη και αυτό είναι απλό γεγονό. δεν είναι κριτική γιατί με βάση τα δεδομένα του 2001 δεν μπορούμε βεβαίως να ξεκινήσουμε έργο. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Κομισιόν και ειδικά για το Fusion for Energy και για τους άλλους συμμετέχοντες να συγκεντρώσουν τα δεδομένα, τα στοιχεία και να υποβάλουν ένα σχέδιο στο οποίο θα λένε ποιο κόστος μας περιμένει στο μέλλον. Ακόμα και αν ξέρω πως δεν είναι απλό να κάνει κανείς προβλέψεις ε, μακροπρόθεσμες, αλλά χρειαζόμαστε αυτά τα στοιχεία. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Πρέπει να σας πω πρώτα απ' όλα ότι εγώ δεν βλέπω με τον ίδιο ενθουσιώδη τρόπο το πρόγραμμα αυτό όσο η κυρία Γκροστέτ, έστω και αν πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε μακρόθωρη πολιτική. Ε, θεωρώ ότι το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο και επίσης ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι έχοντας βγάλει χρήματα ε, από την ε, κλιματική αλλαγή εν μέρη και αρκετά από την γεωργική πολιτική δεν έχουμε λέω καμία διασφάλιση εγγύηση ότι μετά από 2, 3, 4 χρόνια δεν θα χρειαστούμε επιπλέον χρήματα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι πολλές ευρωπαϊκές ενωσιακές πολιτικές πολιτικές χρηματοδοτούν ένα και μόνο πρόγραμμα, το οποίο όμως το χρειαζόμαστε σήμερα, αυτή τη στιγμή. Το χρειάζεται η βιομηχανία μας και από την άλλη πλευρά έχουμε και πολλά προγράμματα τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή για την ενέργεια, για τις κλιματικές αλλαγές, για τη βέλτιστη χρήση των ενεργειακών πόρων κτλ. Και επομένως ε, ε, ελπίζω ότι θα είναι η τελευταία φορά που μας ζητούν ε, μια επιμήκυνση αυτού του είδους. ναι, και κοιτάξτε, η κυρία Γκροστέτα αναφέρθηκε στους εταίρους. Είμαστε εταίροι, αλλά εμείς είμαστε οι μόνοι εταίρους, στους οποίους ζητούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Οι άλλοι συμμετέχουν σε είδος, είναι διαφορετικό. Κύριε Καταρζή, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, αρκετά σημεία θα ήθελα να θίξω. Πρώτον για τον προπολογισμό. Στον προπολογισμό αυτό έγινε λόγο για το κεφάλαιο 2. Πρέπει να σα πω όμω ότι το κεφάλαιο 2 αφορά όλο το γεωργικό τομέα. Είμαστε πολιτικοί. Ε, και θα πρέπει να πάμε στους γεωργούς να τους πούμε ότι ξέρετε κάτι, θα σας πάρουμε 400 εκατομμύρια να το βάλουμε στο, στο πρόγραμμα ε, ITER. Λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε τώρα, δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε. Δεύτερον, προσθέσατε 15 εκατομμύρια ευρώ από την κλιματική αλλαγή ε, ε, σχετικά με προγράμματα μελέτης της ε, της αποτελεσματικότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ε, ναι, και τι θα γίνει δηλαδή. Ε, Κά, κάτι ταχυδακτηλουργικό έγινε για να μπορούν να φύγουν αυτά τα 15 εκατομμύρια. Αναφερθήκατε επίσης και σε 40 εκατομμύρια περίπου τα οποία θα ε, πάρουμε από, από την Euratom τότε. Δηλαδή τι, δεν θα γίνουν τα μελλοντικά προγράμματα σχάσης, εγώ θα ήθελα θα ήθελα κάποιες επιπλέον ε, πληροφορίες για αυτά τα 540, συγγνώμη, 540 εκατομμύρια. Εάν έχετε κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με προγράμματα, ας πούμε το πρόγραμμα σχάσης στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού, να μας τα πείτε. Λοιπόν, επίσης μιλάτε, για, αναφέρεστε τα χρήματα αυτά και μιλάτε για, τον, ε, ε, για την χρηματοδότηση 12-13. Και εγώ σας λέω τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση μετά το 13. Και τελευταία ερώτηση, γιατί και εγώ πήγα στο Κανταρά. Γιατί μάλιστα είναι και η εκλογική μου περιφέρεια. Άρχισαν ε, οι εργασίες. Αυτό μας είπε και ο κύριο Μπρίσκο αλλά έχουν ξεκινήσει απολύτως παράνομα. Δεν έγινε καμία δημόσια έρευνα. Στο έγγραφο λέει η απόφαση της 22ης Ιουνίου επέτρεψε ε, την, ε, την έναρξη εργασιών εγκατάστασης ε, του ΙΤΕΡ. αλλά ο κύριος Σοζάμι Μποτοζούτα το Σεπτέμβρη λέει ότι θα ξεκινήσει στα τέλη τρέχοντος έτους η δημόσια έρευνα. Ναι, αλλά ποιος κροϊδεύει ποιον εδώ. Ξεκινήσατε λοιπόν τις εργασίες, ξεκινήσατε τις κατασκευαστικές εργασίες για να χτίσετε το κτίριο και μετά θα κάνετε την έρευνα. Ε, ε ναι, αλλά τότε ποια αξιοπιστία θα έχετε στα μάτια του τοπικού πληθυσμού. Πρώτα θα έπρεπε να έχει γίνει η μελέτη και η έρευνα και μετά να ξεκινήσουν τα έργα. Επομένως, έχουμε προϋπολογισμό ο οποίος εκρήγνεται ε, γιατί έχει τριπλασιαστεί ανάμεσα στο 2001 και το 2010. Δεύτερον, βρισκόμαστε στην πλήρη παρανομία και τρίτον, βρισκόμαστε σε μια πλήρη αντιδημοκρατική κατάσταση απέναντι στους πολίτες. Ευχαριστώ. Οπωσδήποτε θα απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Κυρία Ντεκαστήγιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους ε, των διαφόρων φορέων για τις εξηγήσεις που μας έδωσαν. Δεν πρόκειται να επαναλάβω πράγματα τα οποία έχουν ήδη υποθεί. Θα ήθελα να ασχοληθώ μονάχα με τις μεγάλες γραμμές ε, του θέματος. Ε, ε, κάνατε μια καλή σύνθεση και εσείς ο ίδιος. Είναι γεγονός ότι αντιμετωπίσαμε ένα μεγάλο πρόβλημα, γενικευμένο πρόβλημα διαχείρισης ε, του έργου. Από την σύλληψη μέχρι διαχείριση των οικονομικών πόρων, των διοικητικών πόρων, του ανθρωπίνου δυναμικού. Υπήρξε πρόβλημα. Αλλά νομίζω στρεφόμενοι και προς το μέλλον ότι είναι πιο σημαντικό να πούμε ότι υπήρξε αποτυχία όσον αφορά τη διαχείριση, δηλαδή το τμήμα της διαχείρισης που έπρεπε να αναγνωρίσει την, διαρκή διολίστηση των στόχων και των κονδυλίων δεν λειτουργήσε. Αυτό το κομμάτι της διαχείρισης δηλαδή απέτυχε πλήρως. τελικά δεν μπορέσαμε να καταφέρουμε να ε, δούμε σαφώς και να ορίσουμε σαφώς ούτε τους στόχους ούτε τα κονδύλια. Θα πρέπει στο μέλλον να υπάρχουν οι μηχανισμοί οι οποίοι θα μας επιτρέπουν να είμαστε σίγουροι ότι στο μέλλον θα πάνε καλά τα πράγματα. Κοιτάξτε, εγώ έχω πλήρη εμπιστοσύνη στο πρόγραμμα, το θέλω το πρόγραμμα, αλλά όπως έλεγαν και κάποιοι συνάδελφοι, ίσως θα πρέπει να ληφθούν κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Εγώ θέλω να ξέρω πάντως το εξή. Σε αυτή τη νέα δομή, σε αυτήν την ε, διαδικασία ε, επαναδιατύπωσης ας πούμε των διαφόρων ε, τομέων διαχείρισης πώς προτίθεστε να, να, διορθώσετε τα προβλήματα και πώς προβλέπετε, ποιος μηχανισμός προβλέπετε έτσι ώστε κάθε φορά που παρουσιάζεται πρόβλημα να προειδοποιήσετε έγκαιρα. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Λοιπόν, θα σταματήσουν τώρα οι ερωτήσει για να απαντήσει ο κύριο Ζανζάν γιατί πρέπει να φύγει και υπάρχουν πολλά σημαντικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν οπωσδήποτε. Οπότε θα ακούσουμε τώρα κάποιε πρώτε απαντήσει. Δεν έχει νόημα να συσσωρεύονται ερωτήσει και να φύγει μετά ο κύριο Ζανζάν. Οπότε, παρακαλώ απαντήστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω στα δημοσιονομικά και θα αφήσω το φίλο και συνάδελφο να απαντήσει στις υπόλοιπε. Για τη χρηματοδότηση. Η προέλευση των κονδυλίων και αναφέρθηκε κυρίως το, ε, σχετικά με το 2 το ερώτημα. Δηλαδή, ε, έχει τα αναγκαία κονδύλια η προσπάθεια αυτή. Όχι. Εδώ έχουμε κονδύλια που δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2010. στη Γεωργία το οικονομικό έτος ολοκληρώθηκε στις 15 Οκτωβρίου. Παρακολουθείτε λοιπόν για κονδύλια, τα οποία είναι διαθέσιμα, που κανονικά επιστρέφονται στα κράτη-μέλη, γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν, ε, οφείλονται στους εθνικούς προϋπολογισμούς και τώρα λέμε, έχουμε ένα περιθώριο εδώ διαθέσιμο από τις ε, αγροτικές δαπάνες και το τραβηχτικό δικαίωμα που διαθέτουμε τα, το μεταφέρουμε στο α, 1α, δηλαδή εκεί που καλύπτονται οι δαπάνες του προγράμματος ΙΤΕΡ. Δηλαδή δεν στερούμε από την Ευρωπαϊκή Γεωργία το παραμικρό. Υπάρχουν πόροι διαθέσιμοι στο εσωτερικό των ε, γραμμών του υπολογισμού του 2010 που δεν είναι πλέον διαθέσιμοι στο τέλος του 2010. Εξού και είναι κάτι να ληφθούν αποφάσεις από αυτού πριν το τέλος του χρόνου, Γάλλους, τα ε, κονδύλια αυτά θα χαθούν από τις ευρωπαϊκές δαπάνες. Πάει αυτό. Θα έλεγα δηλαδή ότι εντός αγωγικών έχουμε μια ευκαιρία που για κάποιους λόγους σε κάποιες ε, αγροτικές δαπάνες ήταν πολύ κάτω από το ανώτατο όριο που είχε προβλεφθεί στον προπολογισμό του 10. Δεύτερον, όσον αφορά τη χρηματοδότηση ε, και την αναδιάταξη. Τα 460 εκατομμύρια. Οι ο συνάδελφος θα σας πει τις λεπτομέρειες του τι μπορεί να γίνει, τα πλαίσια, προγράμματος πλαισίου. Πάντως αυτά τα 460 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το σύνολο του προπολογισμού δεν είναι μεγάλο ποσοστό. Μιλάμε για 2 περίπου της 100 του συνόλου του προπολογισμού. Πρόκειται για μια σημαντική, ε, ένα σημαντικό κονδύλι, αλλά που σχετικά με το διαθέσιμο είναι αρκετά μικρό. Υπάρχει και ένα backloading κάθε χρόνο των δημοσιονομικών προοπτικών του, μέχρι το 2013 κάθε χρόνο έχουμε ε, ένα δισεκατομμύριο διαθέσιμα κονδύλια για τα προγράμματα αυτά. Τρίτο ερώτημα. Τι γίνεται στην πραγματικότητα αν ξεπεραστεί ε, ο προπολογισμό μετά το 2013 δηλαδή. Η, η, η θέση της Κομισιόν είναι πολύ ε, σαφής. Είχε γι' αυτό δυσκολεύτηκε πολύ με τα κράτη-μέλη στη συζήτηση στα συμπεράσματα του Συμβουλίου τον Ιούλιο. Είπε η Κομισιόν ότι δεν τίθεται θέμα, δεν πρόκειται να θυσιαστούν οι άλλες πολιτικές υπέρ Και για να πω τα πράγματα ξεκάθαρα, δηλαδή δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα μειωθούν, θα περιορίσουμε τις φιλοδοξίες μας στους άλλους τομείς και γι' αυτό η διαθεσιμότητα κονδυλίων ε, για τις αγροτικές δαπάνες, απλώς, από τις αγροτικές δαπάνες, απλώς είναι μια καλή ευκαιρία. Αυτό που λέμε, είπαμε και θα συνεχίσουμε να λέμε στα κρατημέλη είναι το εξή. Είμαστε διατεθειμένοι να εισάγουμε κάποια ποσά για τη χρηματοδότηση ε, από τον προϋπολογισμό των μεγάλων έργων. Όμως ο κοινοτικός προϋπολογισμός δεν μπορεί σε μόνιμη βάση να χρηματοδοτεί τις υπερβάσεις. Άρα θα πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αυτό το ζήτημα. Όσον αφορά το πρόβλημα του ΙΤΕΡ, η Κομισιόν ανέφερε ότι η παρέμβαση του κοινοτικού προϋπολογισμού θα σταματήσει στο 1,4 δις για ε, τις συμπληρωματικές δαπάνες και ότι αν υπάρξουν άλλα προβλήματα πλέον θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Στην Budget Review η Κομισιόν ανέφερε ότι ότι συμφωνεί να μελετήσει αν πρέπει να δημιουργηθούν συγκεκριμένες δομές υποδομής ε, μεγάλων προγραμμάτων που θα χρηματοδοτούνται από συγκεκριμένα κονδύλια του προϋπολογισμού. Αυτά είπαμε και αυτά θα λέμε στις προτάσεις στο πλαίσιο της επόμενης ε, χρηματοδοτικής προοπτικής. Αυτά ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε. Θα επαναλάβω και θα επιμείνω την ανάγκη να βρεθεί μια λύση για τη χρηματοδότηση αυτού του 1,4 δις εντός του πλαισίου της διαβούλευσης που θα γίνει μεθαύριο στο Συμβούλιο. Χαίρομαι που ακούω τώρα ότι από πλευρά Συμβουλίου υπάρχει ένα κάποιο άνοιγμα απέναντι στην Κομισιόν. Θυμίζω ότι τον Ιούλιο το Συμβούλιο ήθελε μία πλήρη αναδιάταξη εντός του 1α. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση που αλλάζει αυτή η ακραία θέση του Συμβουλίου και ελπίζω ότι και το Κοινοβούλιο θα στηρίξει την πρόταση της Κομισιόν, η οποία προσπαθεί υπό τις παρούσες συνθήκες να πετύχει κάτι που είναι ε, μοναδικό για την πρόθεση αυτού του έργου του σημαντικού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις σαφείς απαντήσεις σας. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Σμίτση για τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. κάποιες απαντήσεις. Να υπογραμμίσω την εκτίμηση μας για την υποστήριξή σας στο πρόγραμμα ΙΚΑΡ. Ένα πρόγραμμα που δεν είναι δυνατόν να μην φτιάξουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε με αυτή την προσέγγιση. Ιδάλλως, στο μέλλον ε, θα έχουμε προβλήματα στην ε, παροχή ενέργειας και κυρίως όσον αφορά ε, τους ε, περιβαλλοντικούς στόχους για τις εκπομπές διοξίδιου του άνθρακα που έχουμε θέσει. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε, να το διερευνήσουμε αυτό. Και μάλιστα κυρίες και κύριοι μέλη της Επιτροπής πρόκειται για ένα αρκετά επικίνδυνο πρόγραμμα όπως συμβαίνει με όλα τα ερευνητικά προγράμματα αλλά δεν μπορούμε να μην το προχωρήσουμε. Όσον αφορά την... Ε, υπάρχει ένα θέμα αξιοπιστίας, διεθνούς αξιοπιστίας. Αναλάβαμε αυτό το πρόγραμμα, δεσμευτήκαμε, ε, συνεργαζόμαστε με άλλους εταίρους ε, διεθνώς και περιμένουν από εμά να καθοδηγήσουμε. Και αν παρατηθούμε, αν δείξουμε ότι δεν έχουμε αφοσίωση σε αυτό, είναι σοβαρότατο ατόπιμα στη διεθνή αρένα. Ακούσατε ότι πρέπει να βρεθούν τα 1,4 δις όχι όμως σε βάρος του προγράμματος πλαισίου. Αυτό ε, αναφέρθηκε από πολλούς από εσά. Και αυτό το έχουμε πει και εμείς. Το πρόγραμμα πλαίσιο προσφέρει κάτι, εντάξει, λογικό. Και προς το παρόν τα 360 προγράμματα που προέρχονται από το πρόγραμμα πλαίσιο είναι σαφώς λογικό ποσό. Αν θα ξαναγίνει τώρα κάτι τέτοιο. Ω νέο γενικό διευθυντή θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Αυτή η υπέρβαση του κόστου και το διοικητικό πρόβλημα. Γιατί από τότε που ανέλαβα τον Ιούλιο έχω να αντιμετωπίσω αυτό το θέμα και θέλω να το ολοκληρώσω, να το, να το κλείσω. Και έχουμε ήδη λάβει αρκετά δραστικά μέτρα. Άλλαξε η νομή διοίκηση του Διεθνού Οργανισμού ITER και του Fusion for Energy που βρίσκεται στη Βαρκελόνη. Λήφθηκαν οδυνηρέ αλλά απαραίτητε από αποφάσεις για να βγουν και να αναλάβουν τα κατάλληλα άτομα. Δεν είναι άτομα που έχουν καλή πολιτική πορεία, είναι άτομα που είναι σε θέση να ε, διοικούν σύνθετα προγράμματα ε, όπως αυτό. Και ε, ο κύριος που κάθεται δίπλα μου είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα τέτοιων ικανοτήτων. Από εμά λοιπόν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ήδη για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Έχουμε υποβάλει τα μέτρα αυτά ε, στα, με τη μορφή ενός εγγράφου που σας υποβάλαμε χθες, θα το έχετε λάβει σήμερα το πρωί. Ζητώ συγγνώμη που το ε, αργήσαμε. Θα επανέλθω όταν το έχετε μελετήσει για να το συζητήσουμε. Θα ήθελα να ήταν έτοιμο για αυτή τη συνάντηση απλούστατα για να σας δώξω ότι δεν έχουμε έρθει εδώ να ζητήσουμε επιπλέον χρηματοδότηση, αλλά έχουμε έρθει και με λύσεις για να βελτιώσουμε τη διακυβέρνηση και τη διοίκηση τι άλλο που με αναχλονεί και θέλω να σας το ομολογήσω, αλλά δεν αφορά εσάς, είναι τα κράτη, αφορά τα κράτη-μέλη. Χάρη στον κύριο Μπρίσκο έχουμε ήδη κάποιες σοβαρές ε, ε, εξοικονομήσεις, έχουμε πετύχει ε, εξοικονόμηση κονδυλίων και τώρα το Συμβούλιο λέει «Α, ξοδέψατε λιγότερα, άρα δεν θέλετε το 1,4 δις». Δεν είναι ρεαλιστική αυτή η κατάσταση λέμε με τον αριθμό των κρατών μελών θα κάνουμε τα πάντα για να δημιουργήσουμε αποθέματα, να ε, υπάρξουν ε, περικοπές κόστους, να μην έχουμε προβλήματα σε 3-5 χρόνια, να μείνουμε στο 6,6 που είναι το μέγιστο, αλλά βεβαίως γι' αυτό χρειαζόμαστε πλήρη πολιτική στήριξη από εσά στο να δοθούν αυτά τα 1,4 δι τα επόμενα χρόνια. Ιδάλλως, σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να αφήσουμε να ε, διακυβεύεται η διεθνή μας φήμη να καταστραφεί αυτό το έργο και είναι ένα θέμα ασφάλεια που πρέπει να επιδιώξουμε να μην παραιτηθούμε από αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπρίσκο. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, παρακαλώ. Ναι. Ναι, ε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Έγινε μια παρατήρηση για το αν και κατά πόσον είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε ίσως υπήρξε παρεξήγηση. Προσπάθησα ευθύς εξ αρχής να εξηγήσω ότι το ίτερ προχωράει έτσι και αλλιώ. Μπαίνει στη φάση της κατασκευής. Τώρα αν και κατά πόσον είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε πραγματικά. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αποφασίσαμε ε, ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν. Ξεκινήσαμε να τις κάνουμε. Ίσως ε, χρειαστούν έξι και παραπάνω μήνες πριν γίνουν και ολοκληρωθούν, αλλά είμαι βέβαιος ότι προχωρούμε προς σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά το κόστος, ρωτηθήκαμε για τις εγγυήσει και για το να ξανάρθουμε τυχόν. Θα προσπαθήσω να σας ε, ησυχάσω επ' αυτό. Παρότι σε ένα τέτοιο είδου έργο δεν μπορεί πραγματικά να εγγυηθεί κανείς τίποτα. Όμως, εδώ και δύο χρόνια ξεκίνησαν αυτές οι νέες ε, εκτιμήσεις για το κόστος. από τότε, ή μάλλον, πρέπει να πω, ελέγχθηκαν από ομίλους και ομάδες ε, ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων, άρα έχουν κάποια εγγύηση. Αλλά μέσα σε αυτό το διάστημα των δύο ετών δεν είχαμε δυσάρεστες εκπλήξεις. Ζούμε με το, τις εκτιμήσεις αυτές του τότε ενώ στην προηγούμενη διετία τριετία όλο και προέκυπταν εκπλήξεις ε, πράγματα που είχαν ξεφύγει από την αρχική εκτίμηση του κόστους ε, μέχρι στιγμής εμείς τώρα δεν έχουμε άσκημες εκπλήξεις. Τρίτο θέμα σχετικά. Ε, όπως σας είπα, ήδη ε, τα συμβόλαια και παρακολουθούμε ε, τις τιμές που υπάρχουν στη βιομηχανία και πώς συγκρίνονται με τον προπολογισμό του, ε, του κόστους του δικού μας. Μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι θετικά. Οι συμβάσεις που αναθέτουμε είναι μάλλον χαμηλότερες από τους προϋπολογισμούς τους οποίους στηρίχθηκαν οι εκτιμήσεις κόστους που και πάλι δείχνει ότι είναι καλές ε, οι εκτιμήσεις κόστους αλλά και λίγο πιο ψηλά από ότι η πραγματικότητα, αλλά το, υπερ, υπογραμμίζουμε αυτό. Υπάρχει ακόμα αυτό το 6,6. Αυτή τη μείωση την διευθετήσαμε αρκετά απλά ή όταν προτάθηκε με το να σταματήσουμε ε, να, να, διαγράψουμε το αποθεματικό. Είχαμε 160 εκατομμυρίων. Στην ουσία αυτό το αποθεματικό, αυτό το ποσό για έκτακτες ανάγκες το διαγράψαμε. Αυτό τότε ήταν εύκολο και να το κάνουμε και να το πούμε. Οποιουδήποτε όμως τέτοιου εκτάσεως έργου χρειάζεται ένα αποθεματικό εκτάκτου ανάγκης. Και οι αναθέσεις συμβολέων που έγιναν μπορούν εύκολα να τραπούν το επόμενο διάστημα. Έτσι λοιπόν, πέρα από την προσπάθεια περιορισμού του κόστους, πρέπει να ξαναφτιάξουμε ένα τέτοιο αποθεματικό. Αν κάνουμε περικοπές κόστους το επόμενο διάστημα, εγώ φιλοδοξώ να τις ε, μεταφέρω, να μεταφέρω τα ποσά σε ένα τέτοιο αποθεματικό, ώστε να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα χωρίς να χρειαστεί να ξαναστραφούμε σε εσά. Υπήρχε και μια άλλη ε, σχετική ερώτηση όσον αφορά ε, την ε, συστήματα ε, παγρύπνησης κλπ. Αυτό θα απαντηθεί με τις διαδικασίες του project management που δημιουργούμε. Αυτές ε, μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε την πραγματική πρόοδο του έργου. Αν και κατά πόσον μέχρι κάποια στιγμή έχει γίνει αυτό που έχουμε πει ότι θα γίνει και αν έχουμε πληρώσει για αυτό το έργο όσο είχαμε πει ότι θα πληρώσουμε υπάρχουν τυποποιημένες τεχνικές που ε, από εδώ και στο εξή θα εφαρμόζονται και που πρέπει και θα δείξουν ότι δεν θα υπάρξουν περίοδοι κατά τις οποίες δεν θα γνωρίζουμε τι ακριβώς γίνεται. Ε, τέλος, σχετικά με το θέμα ε, ε, τη δουλειά στο Κάνταρας. Δεν αντιμετωπίζουμε τις γαλλικές αρχές, το ΕΦΑΡΗ. E. Αυτό είναι ε, δουλειά του Διεθνούς Οργανισμού στο Κανταράς, αλλά δεν υπάρχει παράνομη κατάσταση. Έχουμε εξάλλου τις ε, άδειες ε, κατασκευής και οικοδομής. Αν χρειαστούν περαιτέρω άδειες, ευχαρίστως να το συζητήσουμε μεταξύ μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λοιπόν. Ο κύριος Οντή κατόπιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτέλους έφτασε το θέμα και στο Κοινοβούλιο. Επιτέλους θα συζητήσουμε μεταξύ Κοινοβουλίου, δηλαδή Συμβουλίου και ε, Κομισιόν. Αρκετές ε, σκέψεις θα κάνω. Μερικές σχετικά με το ίδιο το ίτερ. Πρώτον, λειτουργεί. Η τεχνολογία το ΚΑΜΑΚ δουλεύει σε μικρή κλίμακα. Σε μεγάλη κλίμακα είναι αυτό που βλέπουμε στα αστέρια. Ε, επομένως, ε, λυπάμαι γιατί ενώ έχουμε τόσο καλά στοιχεία όσον αφορά την έρευνα και την επιστήμη, ε, πολύ συχνά μιλάμε μόνο για τα χρήματα και για την δημοσιονομική διάσταση. Επίσης, το πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Ήδη την εποχή του Γκορμπατσέφ η Ρωσία. Ε, η, Βραζιλία ήδη έχει υποβάλει αίτημα συμμετοχής. Ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε. Πρόσφατα έγινε η διάσκεψη κορυφής Ασίας-Ευρώπης. Ούτε λέξη για το πρόγραμμα αυτό. Ούτε ε, ε, καμία αναφορά σε ενδεχόμενο ας πούμε τηλεδιασκέψεων με, ε, με φοιτητές, μελετητές που θα μπορούσαν να μάθουν ένας από τον άλλον σωρό πράγματα. Γιατί δεν ζητάμε και από τους Κινέζους μια τέτοια επαφή. Τέλος, εμείς κάνουμε τη δικιά μας θέση. Η Γεωργία, το PSRD, έχουμε πλεονάσματα κάθε χρόνο. Όταν κάνουμε τους λογαριασμού μας, πάντα μας μένει ένα δις από εδώ, πολλά εκατομμύρια από εκεί. Μας μένουν πέντε δις, τα δίνουμε ξανά στα κράτη-μέλη. Παραμένει πλεόνασμα σε κάθε ε, σημείο του προϋπολογισμού ε, ε, και νομίζω ότι πραγματικά μπορούμε να μιλήσουμε για την χρήση των πλεονασμάτων. Και επίσης η Επιτροπή που δεν είχε δουλέψει καλά από την αρχή βλέπει ε, την ανάγκη πλέον να υπάρξει και ένα τμήμα επενδύσεων. Ε, δηλαδή το το ψηφιακό, τις ε, υποδομές ενέργειας, το διάστημα είναι τομείς στους οποίους μπορεί και πρέπει το ίτερ να επενδύσει. Ο πρόεδρος Μπαρόζο και η Επιτροπή δεν δούλεψαν πάρα πολύ για την ε, οικονομική αυτή επένδυση στις επόμενε δημοσιονομικές προοπτικέ είπατε ότι θα γίνουν προτάσεις. Μα έτσι πρέπει να δουλεύουμε σε τέτοιου είδου ε, ε, προγράμματα που δεν αφορούν ένα, δύο, τρία χρόνια αλλά ξεπερνούν κατά πολύ ε, τις δημοσιονομικέ προοπτικέ πολλών ετών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά ερωτήματα ετέθησαν σχετικά με τον προϋπολογισμό. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής μονάχα. Τίποτα δεν είναι χειρότερο όταν ξεκινάει κανείς ένα πρόγραμμα διαρκώς να δηλητηριάζεται από οικονομικά ε, προβλήματα. Ε, υπάρχουν δύο όροι και προϋποθέσεις ε, για να μπορέσει το Κοινοβούλιο να ενστεριστεί το πρόγραμμα αυτό. Πρώτος όρος η προϋπόθεση. Να υπάρχει χρηματοδότηση συγκεκριμένα για το πρόγραμμα αυτό ε, και να μην χρησιμοποιεί αυτός ο προϋπολογισμός τα αποθεματικά ή τα πλεονάσματα άλλων γραμμών για να δημιουργεί δικό του πλεόνασμα όταν ας πούμε συναντάμε ε, γαλακτοκόμους, ε, παραγωγούς γάλακτος, ε, δεν είναι δυνατόν να τους εξηγήσετε ότι τα ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν τα πλεονάσματα του γεωργικού προϋπολογισμού γιατί θα δοθούν σε κάποιο άλλο, στο Ταμείο Συνοχής, θα δοθούν κάπου αλλού, αλλά ε, ε, θα χρησιμοποιηθούν σε ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο πρέπει να έχει πλεόνασμα. Δεύτερη προϋπόθεση Και βεβαίως ε, ε, για να τελειώσω μάλλον με την προηγούμενη μου τοποθέτηση, το προηγούμενο όρο, είναι ένα πολιτικό ζήτημα και επίσης ε, δεν είναι πρόβλημα που αφορά ένα έτος. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Εάν υπάρχει το τέλος πλεόνασμα, σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιήσαμε καλά τον προϋπολογισμό μας. Χρειαζόμαστε έναν σταθερό πολυετή προϋπολογισμό εάν η Επιτροπή αποφασίσει ότι στόχος θα είναι το 1 δις 400 εκατομμύρια, εντάξει, αλλά βάσει αυτού να δουλέψουμε. Να μην πούμε ότι ε, ναι θα πάρουμε και λίγα χρήματα από εδώ και άλλα λίγα χρήματα από εκεί και μετά α όχι όχι γιατί θα έχουμε και εμείς πλεόνασμα γιατί κάναμε έτσι τον προϋπολογισμό μας. Αυτό δεν γίνεται. Θέλουμε δέσμευση λοιπόν από το Συμβούλιο στην συζήτηση με το Κοινοβούλιο ε, επί του ενδεχομένου η Επιτροπή να μπορέσει να, έχει, να προσφύγει ε, σε ίδιους πόρους και εάν ε, η Επιτροπή θέλει να είναι αξιόπιστη απέναντι στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να μας κάνει προτάσεις που θα μας δίνουν την δυνατότητα να ε, μετράμε το βάρος των ετήσιων προτάσεων και να είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε την καλύτερη δυνατή ε, χρήση των πόρων, των ε, γεωργικών δυνατοτήτων, ε, της πράσινης ενέργειας κτλ. Όλοι οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ινδία, ακόμα και οι Κινέζοι που θέλουν και να μας ξεπεράσουν, επενδύουν σε, σε νέες τεχνολογίες και σε πράσινες τεχνολογίες. Και εμείς προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε το προπολογισμό μας μονάχα για ένα πράγμα. Είδατε τι έγινε και με τον Καλλιλέο Δουλεύουμε τόσα χρόνια και ακόμα δεν έχουμε τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι τουλάχιστον εδώ θα πρέπει να έχουμε καλύτερη διαχείριση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι ένας ε, εργοδότης και ένας επιβλέπων εξαιρετικά αυστηρός. Θα πρέπει να έχει στα χέρια τη συγγραφή υποχρεώσεων και σαν επιβλέπων να την ε, ε, παρακολουθεί με μεγάλη αυστηρότητα. Και εκεί θα έχει τη βοήθεια του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Αυτά ήθελα να πω και ελπίζω να γίνουν γιατί πραγματικά με ενδιαφέρει το πρόγραμμα αυτό και θέλω να πετύχει. Ευχαριστώ κύριο Στόρμσερ. Ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις έχω προς τους κυρίους και μια ερώτηση προς τη Βελγική Προεδρία με την οποία θα ξεκινήσω. Εάν είμαστε σωστά ενημερωμένοι. Υπάρχει συζήτηση στο Συμβούλιο για την νομική βάση του πώς θα γίνει αυτή η οικονομική συμφωνία. Και εμείς είχαμε καταλάβει πως το Συμβούλιο βασίζεται, αρνείται να βασιστεί στην συμφωνία την διοργανική του 2006, αλλά προτιμά το άρθρο 312, δηλαδή υπό ομοφωνία. Θα μπορούσε να μας ενημερώσει η Βελγική Προεδρία για το πού βρισκόμαστε όσον αφορά την νομική βάση. Για το ζήτημα του κόστους. Είπατε πως υπήρξε κάποιο κόστος πρόσφατα. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες για το κόστος λειτουργίας του αντιδραστήρα και το κόστος διάλυσης. Γιατί αυτά ορίστηκαν το 2001, αλλά εγώ θα ήθελα να ξέρω ποιο είναι το κόστος σήμερα. Και όλο το υπόλοιπο κόστος της επένδυσης έχει ξεφύγει εντελώς. Οπότε όμως προξενούσε έκπληξη εάν η εκτιμήσεις του 2001 εξακολουθούν να ισχύουν. Και νομίζω πως και για την Επιτροπή μας και για το Κοινοβούλιο ολόκληρο είναι πάρα πολύ σημαντική η διαφάνεια. Αλλιώς θα κρύβεται νομίζω και πάλι μια τεράστια αύξηση στο, στο κόστος που θα έπρεπε να γνωρίζουμε. Το άλλο θέμα, εσείς λέτε πως το έργο αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Εάν με έχουν ενημερώσει σωστά και μπορείτε να με διορθώσετε, το ίδιο είναι σε μια πρώτη φάση έρευνας. Μετά, με βάση αυτά τα αποτελέσματα, κάποια στιγμή το 2040-45 θα έχουμε έναν αντιδραστήρα επίδειξης που δεν θα είναι στην Ευρώπη, αλλά στην Ιαπωνία, αν με έχουν σωστά ενημερώσει. Και μετά αν είναι επιτυχής ο αντιδραστήρας επίδειξης θα έχουμε κάποιες εμπορικές ε, εφαρμογές. Οπότε ήδη το 2090 ή 2100 και με μεγάλη αισιοδοξία θα κάνουμε να δούμε, μέχρι τότε θα κάνουμε να δούμε κάποια εμπορική εφαρμογή του έργου αυτού. Και ξέροντας αυτό το έργο και για να απαντήσω και στον κύριο Ντί, δεν ξέρω αν με ακούει, εμείς ως πράσινοι είμαστε υπέρ της επιστήμης, αλλά εάν είναι να λύσω μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση και κλιματική κρίση, έχει υπολογίσει κανείς Εάν παίρναμε τα 15 δισεκατομμύρια και τους 3.000 ερευνητές και τα βάζαμε στην ηλιακή ενέργεια, σε αποτελεσματικές ηλεκτρικές μηχανές και ενέργεια σπίτια μηδενικής ενέργειας για να κάναμε κάποια διεθνή έργα, είμαι σίγουρος πως με όλα αυτά θα είχαμε αποτελέσματα πολύ νωρίτερα και πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Με αυτό νομίζω θα έπρεπε να συγκρίνουμε. Και τέλος για τα ευρωομόλογα, Κατρίν, είμαι υπέρ των ευρωομόλογων, αλλά τα ευρωομόλογα είναι ομόλογα. Δηλαδή σημαίνει πως επενδύει η Ευρώπη κάτι εκ των προτέρων, δηλαδή στις υποδομές θα επενδύσουμε σε γραμμές υψηλές στάσεις και θα πάρουμε τα λεφτά μα πίσω ή σε πίστη στεγαστική και θα πάρουμε τα λεφτά μα πίσω. Αλλά ο αντιδραστήρα αυτό είναι μια μαύρη τρύπα. Πετάμε δισεκατομμύρια και ποτέ δεν θα τα πάρουμε πίσω. Μόνο λεφτά βάζουμε. Γιατί δεν υπάρχει κάποια απόδοση. Οπότε είναι τελείω τελείως λάθος. Εάν θέλουμε δηλαδή, να σκοτώσουμε την ιδέα των ευρωομολόγων, μπορώ να σου το πω απλά. Εάν συνδέσετε τη χρηματοδότηση Twitter με τα ευρωομόλογα, θα σκοτώσετε τα ευρωομόλογα. Γιατί τα ευρωομόλογα μπορεί να γίνουν για κάτι το οποίο θα αποδώσει. Ο αντιραστήρας αυτός δεν θα έχει κάποια απόδοση. Γιατί τα, τα λεφτά δεν θα αποδώσουν τίποτα. Εγώ είμαι υπέρ των ευρωομολόγων, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κρίστιαν Έλερ τελευταίος. Θα ήθελα για εμάς, για την Επιτροπή, ξέρω τι, και για τους, τις συζητήσεις που θα γίνουν για τον προϋπολογισμό. Ακούσαμε και φοβήθηκα εδώ πέρα, γιατί θεωρώ πως τα κράτη-μέλη είναι ανεύθυνα συζήτηση, πως η μείωση από 7,2 σε 6,6 δισεκατομμύρια είναι απαραίτητα αποθεματικά που έφυγαν από το έργο. Αυτό δεν είναι καμία εξοικονόμηση, αυτό είναι κόλπο δημοσιονομικό. Δεύτερον, πρέπει να έχουμε κατά νου και δεν θέλω να με παρεξηγήσει εδώ πέρα η κυρία Γκρουστέτ, ε, για το εάν με ενθουσιασμό θέλω να διατηθούν λεφτά, πρέπει να πούμε πως είπαμε σήμερα σαφώς πως με την έγκριση των χρημάτων από την διαδικασία αυτή του προπολογισμού πρέπει να υπάρχει μια σαφή εικόνα για το πώς θα υπάρξει η διαχείριση του σχεδίου αυτού στο μέλλον και η διεθνής δομή του. Γι' αυτό θέλουμε να μας τα πει αυτά γραπτός για τα τα έχουμε και στη συζήτηση για τον προβολισμό. Το τρίτο ερώτημα, Σίσελιτς παρέμεινε αναπάντητο. Μιλήσαμε για τη διαχειριστική δομή του έργου, αλλά τι γίνεται με τη διαχειριστική δομή της, των γενικών διευθύνσεων. Ποιος, με ποιες αρμοδιότητες στο μέλλον θα ασχολείται με αυτό το έργο. Σκέφτεστε να το δώσετε έξω Θέλετε να έχουμε δικές μας δομές. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι οικονομικά έχει ξεφύγει το έργο. Τρίτη διαπίστωση που μου φαίνεται σημαντική είναι πως τώρα υπάρχει ένας διαχωρισμός, ε, μια διάλυση αυτής της ε, εκτελεστικής επιτροπής και να έχουμε ένα διαχειριστικό υποπτικό συμβούλιο και ένα άλλο που θα ασχολείται με τις προμήθειες. Δύσκολο αυτό και σημαντικό για την δομή και νομίζω σημαντικό για την επιτυχία του έργου. Και τρίτο θέμα που θα ήθελα να θέσω έτσι ε, για λόγους καθαρά λογικής έναντι του κλωτούρμες. Γιατί βέβαια πρέπει να το συγκρίνουμε με το κόστος ευκαιρίας, πόσο μα κοστίζει αυτό σε σχέση με τα λεφτά που παίρνουμε από κάπου αλλού. Αυτό μπορεί να γίνει και για τις ανανεώσιμες, γιατί ελπίζουμε το 2050 να έχουμε 50% της ενέργειας. Δεν ξέρουμε τίποτα. Επιδοτούμε τώρα. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Ε, Τοποθετούμε λεφτά για το μέλλον. Είναι νομίζω εξίσου ε, δικαιολογημένο και αυτό όπως και οι ανανεώσιμες. Και τα δύο είναι μια επιταγή για το μέλλον. Γιατί από πλευρά κόστου ευκαιρία ξέρετε πάρα πολύ καλά πώ μπορούμε να λύσουμε το θέμα του κλίματο. Μπορούμε να χτίσουμε πολύ απλά πυρηνικά εργοστάσια. Καμία εκπομπή και κανένα πρόβλημα με επιδοτήσει. Λειτουργούν χωρί επιδοτήσει σε αντίθεση με τις ΑΠΕ. Οπότε δεν είναι πολύ σοβαρή αυτή η συζήτηση. Έχετε δίκιο όμω, πρέπει να σκεφτούμε ποιο είναι το κόστο ευκαιρία εδώ πέρα. Και αυτό είναι το θέμα για τον προπολογισμό. Και θα βρούμε τώρα για μία φορά λύση για τον προπολογισμό, αλλά πολιτικά πρέπει να μας πει η Κομισιόν για το πώς θα χρηματοδοτεί αυτό εκτός του προγράμματος πλαισίου 7. Δεν μπορεί κάθε πρόβλημα που προκύπτει να το χρηματοδοτούμε από το πρόβλημα πλαίσιο 7 ή 8. Για το μέλλον λοιπόν, γι' αυτό είναι το πολιτικό ερώτημα εδώ πέρα, τι θα κάνουμε στο μέλλον με τον προπολογισμό για τα μεγάλα έργα. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα. Θα ήθελα να δώσω καλεσμένους μας ε, τον λόγο. Λοιπόν, ε, τώρα τα πολιτικά δεν θα τα λύσουμε εδώ πέρα. Να ακούσουμε τις ε, απαντήσεις στα ζητήματα τα τεχνικά. Ευχαριστώ. Πράγματι μιλάμε για ένα μακρόπνο έργο. Και όπως είπα έχει και τους κινδύνους του. Αποτελεί όμως μια ευκαιρία την οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αν πιστεύουμε ή σκεπτόμαστε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν τη λύση και θα μας δώσει ενέργεια τα επόμενα έτη, δεν είναι μια σωστή ιδέα. Πιστεύω ότι δεν είναι ρεαλιστικό. Και η εναλλακτική είναι η πυρηνική ε, σχάση ε, για ενώ εκεί υπάρχουν προβλήματα, ενώ η περινική σύνδεξη, ε, το πρόγραμμα ITER, είναι ένας δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε, είναι ένα πεδίο που αξίζει να διερευνήσουμε. Δεύτερον, πρέπει στο μέλλον να αποφύγουμε όταν υπάρχουν τέτοια ευρεία κλίμακα προγράμματα όπως το ITER ή το Galileo, ε, και υπάρχουν υπερβάσεις κόστους, να υπάρχει ένα πρόγραμμα πλαίσιο ή κάποιο άλλο πρόγραμμα που να πληρώσει γι' αυτό. Ένα άλλο θέμα που αναφέρεται στο έγγραφο της Κομισιόν για το προϋπολογισμό προτείνουμε στο μέλλον να υπάρχει ειδικό κονδύλι του προϋπολογισμού, ειδική γραμμή. Και νομίζω στο προϋπολογισμό ΛΕΚ στο μέλλον πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο προϋπολογισμό που θα αφορά αυτά τα μεγάλα προγράμματα και που πρέπει να χρηματοδοτείται και θα υπάρχει μια συγκεκριμένη εισφορά από την κοινότητα και όχι ποσοστό κάποιου συνόλου. Τρίτον, το θέμα της διεθνούς συνεργασίας ετέθη κυρίως σε σχέση με την Κίνα. Έχουμε τεράστιες επαφές με τους διεθνείς μας εταίρους και οπωσδήποτε σκοπεύουμε να κινητοποιήσουμε αυτούς τους διεθνείς εταίρους για να αυξήσουν ε, την αφοσίωσή τους, τη δέσμευσή τους και να κάνουν περισσότερα. Αλλά πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει η ίδια η Ευρώπη πόσο ενδιαφέρεται για αυτό το έργο. Πρέπει γρήγορα να βρούμε μια λύση αυτό το 1,4 δις. Όλοι οι εταίροι μας, συμπεριλαμβανομένων και των Κινέζων, διερωτώνται ενδιαφέρεται πραγματικά η Ευρώπη για το έργο αυτό. Θέλει να συνεχίσει να επενδύει στη σύνδεξη και θέλουμε αυτό το θέμα πρώτα να λύσουμε πριν πάμε στους εταίρους συμπεριλαμβανομένου τη Βραζιλία ζητώντας ε, τους να επιταχύνουν ή να ε, αυξήσουν την πιθανή εμπλοκή του σε αυτή την προσπάθεια. Η διοίκηση όσον αφορά τις ευθύνε εντό τη Κομισιόν εμείς έχουμε στη δική μας Γενική Διεύθυνση μια εξαιρετική ομάδα που ασχολείται με το ίτερ, είναι άνθρωποι ικανοί, ε, διαρκώς ε, φροντίζουμε να έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση, ε, τις πιο πρόσφατες γνώσεις προσλαμβάνουμε νέους. Το ίδιο συμβαίνει και στο Future for Energy. Είμαστε σε στενή επαφή για να εξασφαλίσουμε ότι και εκεί υπάρχουν κατάλληλοι άνθρωποι, κατάλληλες θέσεις. Μπορεί να πεις ίσως και δύο λόγια για αυτό τα μακροπρόθεσμα δημοσιονομικά ζητήματα. Ο κύριος Μπρίσκο θα πάρει το λόγο τώρα και μετά τα υπόλοιπα. Ρωτήσατε για το κόστος λειτουργίας και το κόστος ε, της, ε, του decommissioning. Πράγματι δεν έχει επανεξεταστεί από τότε που πρώτο ε, υπολογίστηκε το 2001. Μπορούμε να ζητήσουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα είναι τα κυμαίνονται τόσο πολύ όσο το κόστος κατασκευής. Αυτό είναι το ε, κειμενόμενο, το επικίνδυνο. Στην αρχή κοιτάμε το κόστος ανθρώπων, το, στη λειτουργία, το κόστος ε, λειτουργίας των μηχανημάτων δεν είναι τόσο απρόβλεπτα. Στη φάση του decommissioning, της ε, διάλυσης, ε, ε, είναι θέμα της διάθεσης των ραδιενεργών αποβλήτων και τα ταφής. Όλα αυτά είχαν στηριχθεί στις τότε τιμές έχουν αλλάξει, μπορούμε να τα επαναμελετήσουμε, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Τώρα, όσον αφορά το λογιστικό κόλπο, όπως λιγόθηκε, το Συμβούλιο επέβαλε αυτά τα τιμία των 600 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά δεν είπε πώς πρέπει να επιτευχθεί. Η δική μου αντίδραση τότε ε, ήταν αυτή. Δηλαδή ο μόνος τρόπος να το βρω ήταν να θυσιάσω ε, το αποθεματικό για έκτακτα κονδύλια ε, και βεβαίως όπως σας είπα αυτό προσπαθούμε να το ξαναστήσουμε. Ο Τόμας είχε μια ερώτηση προς το Συμβούλιο, θα ακούσουμε την απάντηση. Ένα-ένα. Ας ακούσουμε πρώτα την απάντηση. Also, jetzt der Rat. Ευχαριστώ πολύ όσον αφορά το δημοσιονομικό ζήτημα το οποίο ετέθη κυρίως βάσει της νομιοθετικής ε, βάσης, ε, δηλαδή έγινε σύμφωνα με τη Λισαβόνα ή τη διαθεσμική ε, συμφωνία αυτό το θέμα ε, μελετάτε τούτη τη στιγμή από την νομική υπηρεσία του ε, Συμβουλίου. Επίσης μην ξεχνάμε ότι η συνδιαλλαγή, η διαδικασία συνδιαλλαγής ξεκινάει σε δύο μέρες. Ε, δυστυχώς σας απογοητεύω, αλλά δεν έχει ακόμα αποφανθεί η νομική υπηρεσία. Ευχαριστώ πολύ. Όλα... Ποια ήταν η ερώτησή σας? Ε, ήθελα να αναφερθώ στις ε, τις, ε, και αναφέρθηκε προηγουμένως στις συγκεκριμένες εμπορικές ας πούμε συνθήκες. Είπαμε ότι σε μερικά χρόνια θα έχουμε έναν αντιδραστήρα δείγμα. Ναι, το ίτερ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της τήξης και αναφέρεται βεβαίως και στο 2020. Ε, εάν τα πρώτα αποτελέσματα στο τέλος του, ε, της δεκαετίας του 20 εάν είναι καλά, τότε όντως θα προσπαθήσουμε, θα, μπορούσαμε να ξεκινήσουμε ε, την κατασκευή ενός αντιδραστήρα επίδειξης Ε, ας πούμε τις γενικές γραμμές ε, μπορούμε να πούμε ότι περίπου το 2040 ε, θα έχουμε έναν τέτοιο αντιδραστήρα επίδειξης, ένα demo. Και βεβαίως ενδεχομένως θα υπάρξουν και άλλα τέτοια και άλλοι τέτοιοι αντιδραστήρες επίδειξης και άλλα demos από την Κίνα, από την Ρωσία. Ναι, ναι, είναι γεγονός ότι πλησιάζουμε βέβαια στο δεύτερο μισό του αιώνα. Αλλά εμείς ε, Έχουμε και τις ε, μελέτες πολλών εξάρτητων εμπειρογνωμόνων, οικονομολόγων που δείχνουν ότι θα υπάρχουν πολλές εφαρμογές της τεχνολογίας αυτής μέχρι το τέλος του αιώνα. Ε, ωραία, σας ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι η τελευταία φορά βέβαια που θα συζητήσουμε το θέμα αυτό. Ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ε, πάντως στο μέλλον ε, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα ξεκινήσουμε στην ώρα μας αγαπητοί συνάδελφοι γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και τελικά ορίστε φτάνουμε ε, να ζοριζόμαστε χρονικά. Λοιπόν, χάσαμε λίγο χρόνο, τέλος πάντων να ξεκινήσουμε αμέσως στο επόμενο κομμάτι. We want to start so early as possible. If it's... Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ένα άλλο σημαντικό θέμα και καλό είναι όταν καλούμε συναδέλφους και όταν καλούμε ειδικούς και υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν να τους ακούσουν να γίνονται γρήγορα αυτές οι συζητήσεις. Να ευχαριστήσω εδώ πέρα ειδικά τον συνάδελφο Έλερ, ο οποίος έδωσε την αφορμή για τη μήνυ αυτή ακρόαση. Θα παρακαλούσα οι κύριοι που είναι εδώ στο πόντιουμ όσο δυνατόν πιο σύντομα να δίνουν απαντήσεις ε, στα ερωτήματα για τον ρόλο του άνθρακα στο μελλοντικό ενεργειακό μείγμα για να συζητήσουμε και κάποια πράγματα μεταξύ μας. Δεν θα ήθελα να πω τίποτα άλλο για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Νομίζω πως ο πρώτος είναι ο κύριος Πίκατς. Διευθύνων Σύμβουλος της Βάτενφαλ Πολωνίας και επικεφαλής της πλατφόρμας τεχνολογίας καθαρού άνθρακα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίζω και τους ειδικού. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε για το σεμινάριο αυτό. Είναι τιμή μου να είμαι εδώ σήμερα και να σας πω αυτά τα οποία έχω να σας πω. Λοιπόν, θα μιλήσω στα πολωνικά. Szanowni Państwo, w Europie do produkcji energii... Κυρίες και κύριοι, στην ε, Ευρώπη Λοιπόν, ε, ναι. έχουμε πολιτικούς κινδύνους στο θέμα των, ε, των στόχων μας. Έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που αποτελούν, απαιτούν πολλές επιδοτήσεις. Έχουμε ένα σταθερό σύστημα ε, που είναι ασταθές. Η τέταρτη πηγή είναι ο άνθρακας που είναι το αντικείμενο της σημερινής συζήτησης. Είναι ένα καύσιμο που έχει χρησιμοποιηθεί επί εκατοντάδες χρόνια έχουμε διαθέσιμους πόρους να, για άλλα 200 χρόνια. Η, πόλη, η πόρη αυτή του άνθρακα έχουν ε, μέγεθος πολύ μεγαλύτερο από όλων των άλλων πόρων συνολικά. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, ε, η Κίνα και η Ινδία σε μεγάλο βαθμό για την ενέργειά τους εξαρτώνται από τον άργανα. Περίπου 40% της ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο προέρχεται από τον άνθρακα, τον ανθρακίτη και τον λιγνίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό είναι χαμηλότερο, είναι γύρω στο 28% προς το παρόν και σιγά σιγά πέφτει. Όμως ε, πρέπει να σημειωθεί ότι κάποια κράτη-μέλη έχουν μεγάλη εξάρτηση από τον άνθρακα, κυρίως ε, ε, συγκρινόμενα με τα υπόλοιπα. Ο άνθρακας μπορεί να αποτελέσει εξαιρετική πηγή ενέργειας, διότι ως πηγή ενέργειας ο άνθρακας επιτρέπει μια αξιόπιστη παροχή ενέργειας, ε, χρησιμοποιεί μια γνωστή ε, τεχνολογία και η παραγωγή είναι ευέλικτη. Δηλαδή, άλλες λιγότερο ευέλικτες πηγές ενέργειας μπορούν να αναμειχθούν με το, στο σύστημα παραγωγής. Το καύσιμο αυτό μπορεί να αποθηκευτεί μακροπρόθεσμα και είναι ασφαλές. Η καύση του άνθρακα δεν εξαρτάται από τις καιρικέ συνθήκες. Η κατανομή του άνθρακα ανά τον κόσμο είναι επίσης καλή και σε χώρες που είναι πολιτικά σταθερές. Είναι ένα φθηνό καύσιμο που μπορεί και να χρησιμοποιηθεί και θα χρησιμοποιηθεί από όλο τον κόσμο σχεδόν. Εάν σταδιακά μειώσουμε το μερίδιο του άνθρακα στην παραγωγή ενέργειας, τότε οι, πηγές, οι τιμές της ενέργειας στον καταναλωτή θα αυξηθούν η καύση του άνθρακα για την παραγωγή ενέργειας δεν αντιβαίνει τη χρήση πυρηνικής ενέργειας ή ε, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όλες αυτές οι πηγές έχουν τα καλά και τα αρνητικά τους. Χρειαζόμαστε μια σωστή αξιολόγηση και μια, ένα σωστό ενεργειακό μείγμα. μία μονοκαλλιέργεια ανανεώσιμων θα είναι πιο δαπανηρή και λιγότερο ασφαλής. Το, ο άνθρακας είναι υπαρκτός, φθηνός και σταθερός. Έχει ένα αρνητικό την εκπομπή, την παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα. Η Ευρώπη δεσμεύτηκε να μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου ως κομμάτι της αντιμετώπισης του κλιματικής αλλαγής. Όμως χρειαζόμαστε ενέργεια και ε, η ανάγκη, η ζήτηση της ενέργειας θα αυξηθεί. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι ο άνθρακας θα συνεχίζει να παίζει ρόλο. Δηλαδή θα αποτελέσει ε, μέρος του παγκόσμιου ενεργειακού μείγματος στις επόμενες δεκαετίες. Βεβαίως η Ευρώπη θα κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει ότι η καύση του άνθρακα δεν θα αντιβαίνει ε, τις, ε, τους στόχους μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Όσον αφορά τις ενεργειακές πολιτικές και κλιματικές πολιτικές, η Ευρώπη σκοπεύει να αλλάξει, να αντικαταστήσει την παραγωγή από τον άνθρακα με ανανεώσιμες. Δηλαδή αρχίζουν και παγώνουν οι μονάδες παραγωγής που χρησιμοποιούν άνθρακα. Αλλά θεωρώ ότι η έλλειψη αυτών των μονάδων παραγωγής ενέργειας θα μειώσει τη σταθερότητα της παροχής ενέργειας στην Ευρώπη. Γιατί αν εξαιρέσουμε την πυρηνική ενέργεια και την ενέργεια που προέρχεται από άνθρακα δεν έχουμε άλλες σταθερές πηγές παραγωγής ενέργειας. το πρόβλημα για το περιβάλλον δεν είναι ο άνθρακας, είναι το διοξίδιο του άνθρακα, δηλαδή πρέπει οι εκπομπές να περιοριστούν. Είναι δυνατόν να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της ενέργειας με την ανάμειξη βιομάσας με τον άνθρακα και την συμπαραγωγή ή με τη χρήση της τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης, της CCS. Θέλω να εξετάσω και αυτές τις εναλλακτικές. Συνήθως η παραγωγή από τον άνθρακα έχει ε, αποδοτικότητα μόνο 33%, δηλαδή μόνο το 1 τρίτο ε, παράγει ενέργεια και βεβαίως οι καταναλωτές λόγω των απολειών κατά τη μετάδοση παίρνουν ακόμα λιγότερο ποσοστό. Οι σύγχρονοι οι σύγχρονες μονάδες έχουν ποσοστά παραγωγή 43% για το λιγνίτη και 46% για τον ανθρακίτη. Αν θέλουμε να, αντικατα... αν αντικαταστήσουμε τους παλαιούς από τους νέους σταθμούς παραγωγής ενέργειας θα ε, έχουμε ένα τρίτο λιγότερη απώλεια και θα έχουμε λιγότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Συνεχώς οι επιστήμονες δουλεύουν για την αύξηση της παραγωγικότητας, της ε, αποτελεσματικότητας της παραγωγής ε, των μονάδων αυτών. Επίσης αναφέρθηκα στην συμπαραγωγή ε, ε, ε, με χρήση άνθρακα και βιομάζας που αυξάνει κατά μεγάλο ποσοστό την αποδοτικότητα. Αυτό έχει μια μεγάλη, προσφέρει μεγάλες δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας ταυτόχρονα και το συνολικό, το συνολικό ποσοστό αποδοτικότητας είναι 90% στο χρόνο και ε, παράγονται 140 νομίζω τεραβάτ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό καλύπτει τις ανάγκες μιας ευρωπαϊκής χώρας μεγέθους Αυστρίας. Η τεχνολογία CCS, δηλαδή δέσμευσης και αποθήκευσης, είναι ένας άλλος τρόπος μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή εδώ συλλέγονται το 90% των εκπομπών από του συμβατικού σταθμού ε, όπως γνωρίζετε, η τεχνολογία CCS έχει δοκιμαστεί στον πετροχημικό κλάδο, ας πούμε. Το πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα ε, δέσμευσης του άνθρακα ήδη λειτουργεί. Η, η αποθήκευση σαφώς ε, λειτουργεί και είναι ασφαλής η τεχνολογική αυτή εξέλιξη του CCS είναι χαρακτηριστική οδός ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, οι οποίες θα πρέπει να μπουν στην εμπορική φάση. Η ενδιάμεση φάση που είναι ενώ ε, ακόμα το μέλλον ε, είναι η δημιουργία ε, μονάδων επίδειξης, τα demo. Έχει έχουν γίνει ρυθμίσεις ε, για τη λειτουργία αυτών των μονάδων επίδειξης που σκοπό έχουν τη βιωσιμότητα της τεχνολογίας αυτής. Όμως η πρόοδος είναι αρκετά βραδιά, βραδία. Μοιάζει ε, να βραδιπορούμε, οι επενδύσει τές δεν μιλάνε πλέον για κατασκευή ε, μονάδων επίδειξης CCS, μιλάνε για ότι επιθυμούν και σκοπεύουν να φτιάξουν τέτοιες μονάδες αν υπάρξουν οι σωστοί κρατικοί κανονισμοί, αν υπάρξει οικονομική στήριξη και αν τα σχέδια γίνουν αποδεκτά από την κοινωνία. Ένα ασταθές ρυθμιστικό πλαίσιο, η οικονομική κρίση καθώς και η έλλειψη δημοτικότητας, η περιορισμένη δημοτικότητα αυτών των ε, ε, επενδύσεων σε υποδομές ε, έχει οδηγήσει σε δραστικό περιορισμό των επενδύσεων σε αυτό το κλάδο. Δηλαδή το έργο CCS έχει ε, πληγεί από αυτή την εξέλιξη ως αποτέλεσμα μπορεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να οδηγηθούμε σε αστάθεια της ασφάλειας της παροχής ενέργειας. Επίσης μπορεί να δυσκολευτούμε να πετύχουμε τους στόχους μας για το κλίμα. Αν δεν προχωρήσει το CCS και το περιορισμό του κόστους τους, πολύ λίγε θα είναι οι χώρε που θα χρησιμοποιήσουν αυτή την τεχνολογία γι' αυτό. Οι επιχειρήσει παραγωγή ηλεκτρισμού που θέλουν να ε, υιοθετήσουν το CCS θα πρέπει να ενισχυθούν. χωρί αυτή την υποστήριξη η τεχνολογία αυτή δεν θα εισαχθεί στον ενεργειακό τομέα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Απο, απαιτείται πολιτική στήριξη. Η ασφάλεια τη παροχή ενέργεια απασχολεί και του καταναλωτέ και τι επιχειρήσει τη Ευρωπαϊκή. Ευρώπης. Δεν είναι θέμα απλώς και μόνο για τον ενεργειακό κλάδο. Είναι πρόκληση και για τους νομοθέτες αλλά συνολικά και για την κοινωνία. Αν αφήσουμε τις ε, εταιρείε ενέργειας ε, χωρίς βοήθεια το αποτέλεσμα θα είναι ελλείψεις σε αυτό το τομέα σε διάφορες χώρες η ανάπτυξη, η πρόθεση του CCS είναι ένας τρόπος να περιοριστούν οι εκπομπές σε τρίτες χώρες. Οι επιχειρήσεις ενέργειας μπορεί να αποτελέσουν τους πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ένωσης αλλά δεν μπορούν από μόνες τους να αναπτύξουν μια τεχνολογία που σε μεγάλο βαθμό θα χρησιμοποιηθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης δεν πρέπει να τις εγκαταλείψουμε όσον αφορά το να πιστεί ο κόσμος ότι αυτή η τεχνολογία είναι αποδεκτή. Οι κυβερνήσεις και άλλες αρχές μπορούν να παίξουν τεράστιο ρόλο σχετικά. Εν κατακλείδη μπορώ να πω ότι το, ο άνθρακας μπορεί και πρέπει να γίνει στο μέλλον σημαντικό συστατικό του ενεργειακού μείγματος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει όμως να είναι το είδος του άνθρακα που δεν θα εκπέμπει διοξίδιο. Αν δεν εκπέμπει διοξίδιο ο άνθρακας θα πρέπει να ε, έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κλάτη μέλη. Η στήριξη πρέπει να δοθεί και στις μονάδες επίδειξης, πρέπει να οικοδομηθούν γρήγορα χώρα μέσα χρηματική στήριξη. Φοβάμαι ότι η φυστάμενη στήριξη είναι ανεπαρκής. Οι επιχειρήσει ενέργειας δεν πρόκειται από μόνες τους να αναλάβουν αυτό το κόστος. Ε, μπορούν να καλύψουν κάποιο από το, ένα μέρος του κόστους κατασκευής, αλλά όχι να τον αλάβουν εξ ολοκλήρου. Οι κυβερνήσεις πρέπει να ε, προωθήσουν την απαραίτητη νομοθεσία ε, για το CCS χωρίς να βάλουν υπερβολικά το βάρος της επιχειρήσεις ενέργειας και θα πρέπει να ενθαρρύνουν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, να ενθαρρύνουν τον πληθυσμό να δεχτεί ε, περισσότερο αυτή την τεχνολογία. Ιδάλλως, την επόμενα 20 ή 30 χρόνια θα μιλάμε για έναν ε, ενεργειακό τομέα στην Ευρώπη χωρίς άνθρακα, αλλά τότε θα έχουμε την ακριβότερη ηλεκτρική ενέργεια στον κόσμο. Αν δεν καταφέρουμε να καταδείξουμε ότι το CCS είναι ανταγωνιστική τεχνολογία, αν δεν καταφέρουμε να καταδείξουμε ότι η κάψη του άνθρακα και η μείωση του διοξίδιου του άνθρακα μπορούν να προχωρήσουν παράλληλα, τότε οι ελπίδες μας για μείωση των ε, παγκοσμίων εκπομπών θα χαθούν. Η καύση του άνθρακα έχει λαμπρό μέλλον και πρέπει να αποφασίσουμε πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτό. Ευχαριστώ. Κατόπιν θα δώσω τον λόγο στον κύριο Πόλα Αλόνζο, Γενικό Διευθυντή Ορυχείων και Ενέργειας στο Περιφερειακό Υπουργείο Βιομηχανίας του Πριγκιπάτου της Αστουρίας. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την Ευρωπαϊκή, την, συγγνώμη, την Επιτροπή Έρευνας που με προσκάλεσε σε αυτήν την ε, συζήτηση ε, για να συζητήσουμε για το θέμα του άνθρακα ε, στα πλαίσια του νέου ενεργειακού μείγματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την Ισπανία και για την Αστούρια συγκεκριμένα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δούμε, να κάνουμε μία σύνοψη της της παρούσας κατάστασης καθώς επίσης ε, και του μέλλοντος που θέλουμε να έχουμε τα επόμενα χρόνια. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε ότι η Ευρώπη εξαρτάται πάρα πολύ από το ε, εξωτερικό όσον αφορά ε, τα ενεργειακά θέματα. Η Ισπανία δε ακόμα περισσότερο. Ε, και ε, παρόλο που η Αστούρια έχει κάποια ανεξαρτησία, παρόλα αυτά δεν καταφέρνουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Έχουμε μεγάλη λοιπόν εξάρτηση από το ε, εξωτερικό. Επίσης ε, πρέπει να πω ότι η κύρια ε, χρήση κατανάλωση γίνεται από τις μεταφορές οι οποίες προκαλούν και την μεγαλύτερη μόλυνση άλλωστε. Επίσης δεν υπάρχει αρκετή διασύνδεση ανάμεσα στην ενεργειακή υποδομή ε, της ε, Ευρώπης. Ε, αυτό το στοιχείο γίνεται ακόμα πιο δύσκολο σε χώρες όπως η Ισπανία. Η Ισπανία λοιπόν είναι κατά κάποιο τρόπο ενεργειακά απομονωμένη και επομένως η διασύνδεση με το υπόλοιπο ε, με την υπόλοιπη ευρωπαϊκή υποδομή ενέργειας είναι πάρα πολύ μικρή. Ε, όσον αφορά τώρα ε, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο μείγμα της κάθε χώρας και ακόμα και στην ίδια τη χώρα μπορεί να υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Στην Ισπανία Ας πούμε, ε, είχαμε 16% ε, χρήση άνθρακα και 73% στην Αστούρια. Οι διαφορές μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλες από περιοχή σε περιοχή. Επομένως, χρειάζονται κάποιες κοινέ αρχές. Ε, η τεχνική αηφορία, η οικονομική αηφορία και η ανταγωνιστικότητα, καθώς επίσης και η υπερβολοντική αηφορία. Ε, ο άνθρακας ε, για να μπορέσει να συνεχίσει να χρησιμοποιείται θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να λειτουργήσει καλύτερα. Επίσης έχουμε και πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες ούτε χρησιμοποιούνται ούτε μελετώνται με τον σωστό τρόπο. Ε, ε, εδώ λοιπόν θα πρέπει να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις, ε, να δημιουργηθούν λοιπόν νέες ενεργειακές υποδομές, να υπάρξει διασύνδεση των δικτύων και οπωσδήποτε κάποιες τεχνολογίες υποστήριξης οι οποίες θα επιτρέψουν την καλύτερη διαχείριση της ενέργειας και καλύτερη ενσωμάτωση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οπωσδήποτε εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η έρευνα γενικότερα θα πρέπει να στηριχτεί η καινοτομία ε, κτλ. Και μάλιστα η χρήση της καινοτομίας ε, και στις μεταφορές και σε άλλους ε, τομείς. Έτσι ώστε να έχουμε όσο γίνεται καλύτερη γενικότερη ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Θα σας πω πολύ σχηματικά τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή όσον αφορά το ενεργειακό μείγμα λαμβάνοντα υπόψη τι γενικέ κατευθύνσει γραμμέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και λαμβάνοντα υπόψη την παρούσα κατάσταση, όλε οι ενεργειακέ πολιτικέ ε, στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνηση ε, βασίζονται σε δύο γραμμέ δράση. Ενίσχυση των και ενθάρρυνση των ε, εναλλακτικών μορφών ενέργεια και ενεργειακέ εξοικονομήσει. Βεβαίω, έχουν ληφθεί και μέτρα για την ανάπτυξη δικτύων και διασύνδεσης των ε, δικτύων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την, ε, ε, ε, το εύρος του προβλήματος δημιουργώντας ένα ταμείο για τα θέματα αυτά. Όσον αφορά τώρα την περιβαλλοντική εφορία, αυτός είναι ένας στόχος που στον ενεργειακό κλάδο είχε σαν, έχει σαν στόχο την μείωση των ορυκτών καυσίμων, όσο γίνεται περισσότερο την μείωση των ε, μολυντικών ε, ε, ουσιών και βεβαίως να χρησιμοποιήσει όσο γίνεται περισσότερο το σύστημα παγίδευσης και αποθήκευσης άνθρακας. Ε, βεβαίως αναγνωρίζουν όλοι ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση ο άνθρακας είναι πάρα πολύ σημαντικός και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο όσον αφορά την ενεργειακή ε, την ενεργειακή ασφάλεια της ε, Ευρώπης και αυτό αναφέρεται και στην ε, Πράσινη Βίβλο και στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την δεύτερη ε, για τη δεύτερη ανάγνωση της, ε, της ε, ενεργειακής στρατηγικής. Αναφέρεται επίσης και στην Οδηγία 72 του 2009 και στην Ανακοίνωση Επιτροπής Ε, αηφόρα ε, δημιουργία ενέργειας ε, από, ορικτές, ορυκτά καύσιμα, στόχευση των μηδενικών εκπομπών από άνθρακα μετά το 2020 και κανονισμός του Συμβουλίου 1407 του 2002. Πέρα από τους κατευθυντήριε γραμμέ και του προσανατολισμούς τη Ευρωπαϊκής Ένωση υπάρχουν ε, και μία σειρά μέτρων και ε, δράσεων που έχουν ληφθεί ε, κυρίως από τον τομέα των ορυκτών και επίσης έχουν γίνει και επενδύσεις στι υποδομές των ορυχείων έτσι ώστε να υπάρχουν καλά ικανοποιητικά στρατηγικά αποθέματα ε, άνθρακα ε, και βεβαίως έτσι ώστε να είναι καλύτερη η απόδοση ε, των θερμικών μονάδων καθώς επίσης και των μονάδων Προγέκτος de captura y almacenamiento de CO2. En este sentido... και φυσικά έχουν χρηματοδοτηθεί και μέτρα για την παγίδευση και αποθήκευση ε, του άνθρακα. Στην Ισπανία ε, χρησιμοποιείται ε, και χρησιμοποιούνται και οι εναλλακτικές τεχνολογίες. Ας πούμε η EcoGas χρησιμοποιεί έναν κύκλο με χρήση διάφορων υλικών, εναλλακτικό κύκλο, επίσης ε, σε διαδικασίες προκαύσης ε, και αντίστοιχες, ε, χρησιμοποιούνται, αντίστοιχες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται και στην Περέδα στην Αστούρια. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια χρήσης προφημένων νέων τεχνολογιών ε, αλλά βεβαίως ε, τα αποτελέσματα ε, θα μπορέσουν να καταγραφούν καλύτερα μέχρι το 2020. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στον παρόντο ρόλο του άνθρακα και τον ρόλο του στο παρόν ενεργειακό μείγμα αλλά και στο μελλοντικό ενεργειακό μείγμα. Πρώτα απ' όλα ο ρόλος ε, του άνθρακα ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε τρίτες χώρες ποικίλει. Υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν δικιά τους παραγωγή άνθρακα, άλλες έχουν πολύ αναπτυγμένο τομέα του άνθρακα, άλλες εισάγουν πολύ και άλλες χώρες όπως η Ισπανία έχουν ένα τμήμα παραγωγής μάλλον ήπιο, 10 με 40% και συμμετοχή στο ενεργειακό μείγμα. Μέσω, των, ε, ε, μέσω του νομοθετικού της ε, πλαισίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τον άνθρακα σαν μια πραγματική ε, σαν ένα πραγματικό ενεργειακό πόρο που πρέπει να συμβάλλει στις ε, στα στρατηγικά αποθέματα ενέργειας. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει κυρίως να τονίσουμε την ελάχιστη, την ελάχιστη εγχώρια παραγωγή ε, και την αποθήκευση σε ικανοποιητικό βαθμό έτσι ώστε ε, σε περίπτωση ενεργειακού προβλήματος ή ενεργειακής έλλειψης να μπορεί κανείς να αντιλήσει ε, καύσιμα από την ενέργεια, από, την, το αποθηκευμένο υλικό. Ε, βεβαίως θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι τεχνολογικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά προχωρημένη ας πούμε στην ε, Ισπανία εμείς ε, βασιστήκαμε πολύ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λέμε ότι μέχρι το 2020 43 ε, μάλιστα της της ενέργειας θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και θα στηρίζεται απλώς από τον ε, άνθρακα ε, με εθνική παραγωγή άνθρακα η οποία θα επιτρέπει ε, την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Θα πρέπει να διατηρηθεί η σημασία του άνθρακα στο μελλοντικό ενεργειακό μείγμα και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί ταυτόχρονα με άλλα ερωτήματα δηλαδή την ενεργειακή αποτελεσματικότητα του άνθρακα αλλά και την περιβαλλοντική του επίπτωση ε, είδαμε ότι γίνεται μια προσπάθεια να μειωθούν όσο γίνεται περισσότερο ε, οι εκπομπές. Επίσης ε, η αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα εγώ να υπογραμμίσω τον σημαντικό ρόλο που παίζει στην εθνική ενεργειακή πολιτική κάθε χώρας ο άνθρακας σαν, σαν αποθεματικό ενέργειας. από το, το 1970 μέχρι το 2050 ε, αυξήθηκε η παραγωγή ενέργειας που βασίζεται στον ε, άνθρακα από 40-53% ε, και επομένως ο άνθρακας έγινε πλέον στρατηγικό απόθεμα. έχει οριστεί η ελάχιστο, ελάχιστος όγκος ε, και το ελάχιστο μέγεθος ε, των ε, μονάδων και λήφθησαν και πολύ σημαντικά μέτρα, μέτρα κλειδιά έτσι ώστε να υπάρξει αποτελεσματική αποτελεσματικότητα συγγνώμη, και παρακολούθηση των μονάδων παραγωγής. Ε, θέλουμε, ε, και θέλω να το τονίσω αυτό, ε, να έχουμε competitive mining, δηλαδή έναν ανταγωνιστικό κλάδο εξόριξης. Βεβαίως και το φυσικό αέριο έχει, παρουσιάζει πολύ σημαντικά πλέον εκτήματα το κόστος ε, του άνθρακα ε, ε, ανεβαίνει λόγω του κόστους εξόρυξης και εκμετάλλευσης. Βεβαίως έχουν ληφθεί και πάρα πολλά μέτρα όσον αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Τώρα θα ήθελα να ασχοληθώ με κάποια τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά στοιχεία και τελικά κάποια κοινωνικά και εδαφικά στοιχεία οποία μας οδηγούν στην στήριξη που αποφασίσαμε να δώσουμε στον τομέα του άνθρακα. Θα ήθελα να επιμείνω ε, για μία ακόμα φορά στην ιδέα ε, του καθαρού άνθρακα, ε, του άνθρακα που παίζει σημαντικό ρόλο και που θεωρείται στρατηγικό απόθεμα. Καθαρές λοιπόν μορφές ενέργειας είναι ένα ε, σημαντικό θέμα και για την Ισπανία αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, γενικότερα. Ε, νομίζουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον άνθρακα με καλό τρόπο. 40% έχουμε άνθρακα που παράγεται στην χώρα μας και 60% προέρχεται από εισαγωγές. Βεβαίως το οικονομικό κόστος πρέπει να σας πω ότι είναι μικρό σε σχέση με την επιστροφή ε, και τα κέρδη που θα έχουμε από την καλύτερη χρήση του άνθρακα στο μέλλον. Επίσης, το σύστημα της ε, φορολογίας ε, θα πρέπει να είναι ένα σύστημα φορολογικό το οποίο ε, να δίνει περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης στον τομέα. Βεβαίως, όπως είπα και προηγουμένως, θα πρέπει να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο οι τεχνικές και οι τεχνολογίες παγίδευσης και αποθήκευσης του άνθρακα τα τελευταία χρόνια υπήρξε ε, μια διόρθωση ε, στον ε, κλάδο, αλλά είχαμε επιβάρυνση του κλάδου της εξόριξης. Ανέφερα και προηγουμένως μία σειρά στοιχείων που στο μέλλον θα πρέπει να εξελιχθούν ακόμα περισσότερο τα συστήματα εξόριξης, τα συστήματα καθαρού, ε, καθαρισμού του άνθρακα, καλύτερα συστήματα ε, παγίδευσης αποθήκευση ε, του άνθρακα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ο, ο άνθρακας θα πρέπει να εξακολουθήσει να παίζει ρόλο στον, στο μελλοντικό μείγμα, ενεργειακό μείγμα, γιατί πρόκειται για μια μορφή ενέργειας ασφαλή, η οποία μπορεί να μας βοηθήσει και στο μέλλον πρέπει να αναπτυχθούν βεβαίως ε, κάποιες ε, ε, τεχνολογίες ακόμα περισσότερο έτσι ώστε να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε με όσο γίνεται περισσότερη ανάπτυξη. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία τοπικής ανάπτυξης που συνδέονται με τον άνθρακα και δεν μπορούμε να τα παραμελούμε. Τώρα... Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Νάιτζελ Γκέξλεϊ, πρόεδρο της Eurocoal. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ρόιλ. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι βουλευτέ, κυρίες και κύριοι. Ελπίζω να φανούν οι διαφάνειες λίγο στην οθόνη για να μπορέσετε να δείτε και όλα αυτά όσα θα σας πω. Sorry, it's not me that's being defeated by the technology. These were supplied last week. And... Συγγνώμη, είχα δώσει τις διαφάνειες την προηγούμενη εβδομάδα και περίμενα πως είχε κανονιστεί. Mr. Chairman, would you like to perhaps take some questions while things are sorted out here? Or... Ε, κύριε Πρόεδρε, θέλετε να δεχτείτε ερωτήσεις ή να περιμένουμε να εμφανιστούν οι διαφάνειες. Sorry about this, ladies and gentlemen. What I'm giving you here is a foretaste of the world without technology. Perhaps after that we'll have a world without electricity. Λοιπόν, δεν ξέρω. Ίσως να καταλήξουμε και σε έναν κόσμο χωρίς ηλεκτρισμό. Κάτι το οποίο βεβαίως θα γίνει αν δεν έχουμε άνθρακα. Θα έρθουμε, θα έρθουμε σε σε λίγο σε αυτό. Πριν ξεκινήσουν οι διαφάνειες, ε, να εξηγήσω λίγο πως ε, εκπροσωπώ την Eurocoal, την Ευρωπαϊκή Ένωση Άνθρακα και Λιγνίτη. Είμαι μέλος της Eurocoal, εκπροσωπώ την δική μου οργάνωση, δηλαδή την Ένωση Εισαγωγέων Άνθρακα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πριν από αυτό, Δούλευα βεβαίω ε, στη... στον τομέα των ανθρακοριχείων του Ηνωμένου Βασιλείου. Φαίνεται πως εγώ τώρα μπορώ να δω τις διαφάνειες, αλλά όχι εσείς. Το καλύτερο λοιπόν το οποίο έχω να κάνω είναι να συνεχίσω και να προσπαθήσω να τα πω γιατί εντάξει, οι διαφάνειες είναι για αυτούς που δεν είναι πολύ καλοί ομιλητές και καρτάνε και το κοινό. Ξύπνιο, σαν ελπίζω να τα καταφέρω να μην κοιμηθείτε και χωρίς αυτές. Τι σκόπευα να κάνω λοιπόν σύντομα είναι να θέσω τρία ρητορικά ερωτήματα. Το πρώτο. Εάν ο άνθρακας είναι καύσιμο του μέλλοντος. Και αυτό βεβαίω τίθεται στο παγκόσμιο πλαίσιο και γιατί αυξάνεται και θα αυξάνεται η χρήση του ανεξαρτήτως τι θα συμβεί στην Ευρώπη. Το δεύτερο ερώτημα είναι ένα ζήτημα κλειδί. Εάν ο άνθρακας μπορεί να είναι καθαρός. Εάν η απάντηση ήταν όχι, τότε νομίζω πως ο κόσμος έχει πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Το τρίτο ερώτημα είναι εάν η Ευρώπη χρειάζεται άνθρακα. Και ε, νομίζω πως αυτό το ερώτημα έχει και κάτι παρεπόμενο. Δηλαδή, εάν θα συνεχίσει να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που της δίνει ο άνθρακας. Εάν μπορούσατε να δείτε την επόμενη διαφάνεια θα βλέπατε μία φωτογραφία ενός ε, πολύ μεγάλου και ψηλού στρώματος άνθρακα, γεωλογικού στρώματος, κατά μαύρο, πιο μαύρο και από τις οθόνες που βλέπετε με ύψος 20 μέτρων και πάνω από τα 20 μέτρα υπάρχει γαλανός ουρανός γιατί βρίσκεται βεβαίως στις ΙΠΑ αυτό το ανθρακοριχείο, το στρώμα άνθρακο. Δύσκολο να το φανταστείτε για όσους από εμά γνωρίζουμε βεβαίως τα ορυχεία στην Ευρώπη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ορυχεία άνθρακα, λατομία θα έλεγα, ε, από όπου βγάζουμε πέντε, έχουμε ένα στρώμα 5 μέτρων άνθρακα, το οποίο βέβαια δεν συγκρίνεται με τα 20 μέτρα που θα βλέπατε στην εικόνα. Λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλα τα αποθέματα, μιλάμε για 997 δισεκατομμύρια τόνων ή αρκούν για τις ενεργειακές ανάγκες 144 ετών. Για αποθέματα μιλάμε δηλαδή άνθρακας ο οποίος συμφέρει να εξοριχθεί. Πέραν από αυτά τα αποθέματα υπάρχουν πολλά 3 εκατομμύρια τόνοι πόρων. Οπότε δεν θα τελειώσει το κάρβουνο σύντομα. Και πολλές χώρες που έχουν άνθρακα θα συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν. Το άνθρακα αυτό είναι πολύ διαδεδομένο. Ο άνθρακας αυτός είναι ε, πολύ διαδεδομένος ε, στην Αυστραλία, στην Κίνα, στη Μογγολία, Ρωσία, Καζακστάν, Ουκρανία, Μοζαμβίκη, Νότια Αφρική, Κολομβία και αλλού. Και βεβαίως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αχα. Τώρα θα δούμε. Για το αν σας περιέγραψα σωστά αυτό το οποίο σας είπα, βλέπετε ένα τείχος άνθρακα και βλέπετε και ένα πολύ μικρό όχημα εκεί στο βάθος. Με συγχωρείτε κυρίε και κύριοι. Το είδατε έστω και για λίγο. Λοιπόν, ε, το νόημα αυτής τη διαφάνειας είναι να σας πω πως ο άνθρακας αυτός θα χρησιμοποιηθεί. Οι αναψώμενες χώρες το χρησιμοποιούν και θα βασιστούν στον άνθρακα για την οικονομία τους. Κατά βάση λοιπόν Ah, there we are again. Thank you very much. I think the best thing we can do now. Splendid. Right. So, moving on. Έξοχα. Λοιπόν, παρακάτω. Ο κύριος Πίκατς ανέφερε τις ποσότητες και το ποσοστό άνθρακα που χρησιμοποιείται ανά τον κόσμο, οπότε δεν θα επιμείνω πολύ σε αυτή τη διαφάνεια. Βλέπετε εδώ πέρα κάποια διαγράμματα που μας δείχνουν το ποσοστό άνθρακα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρισμού στον κόσμο, το μεγάλο διάγραμμα, και στην Ευρώπη, το μικρό διάγραμμα. Ίσως είναι πολύ μικρό, δεν το διακρίνεται. Παγκοσμίω, πέραν του ότι είναι το 27% της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας, είναι και το 41% της παραγωγής ενέργειας. Στην Ευρώπη είναι μικρότερο το ποσοστό, είναι γύρω στο 28% και ο λόγος είναι το πολύ μεγάλο κομμάτι της πυρηνικής ενέργειας, πολύ μεγαλύτερο από ό,τι αλλού στον κόσμο. Και αναφέρθηκε και από τον κύριο Πίκατς πως βεβαίως αυτά τα ποσοστά διαφέρουν κατά πολύ ε, στην κάθε χώρα. Παρακάτω ο άνθρακα στην Κίνα. Νομίζω πως μια παρουσίαση για τον άνθρακα δεν θα ήταν πλήρης χωρίς λίγα λόγια για την Κίνα. Η κόκκινη γραμμή που διακρίνεται μας δείχνει την ανάπτυξη κατανάλωσης άνθρακα στην Κίνα που αυξήθηκε πάρα πολύ μετά το 2001 όταν μπήκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου η Κίνα. Είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε όλοι, αλλά νομίζω πρέπει να το τονίσουμε ξανά και ξανά. Η Κίνα ε, εκπροσωπεί το 45% της παγκόσμιας παραγωγής και κατανάλωσης άνθρακα. Αυτή την αλλαγή δεν νομίζω να την έχουμε αντιληφθεί πλήρως, αλλά όλοι βεβαίως ε, απολαμβάνουμε τα αγαθά τα οποία εξάγει η Κίνα. 40 εκατομμύρια iPhone μόνο πέρσι και όλη η παραγωγή τους βεβαίως βασίζεται σε κομμάτια άνθρακα στην Κίνα. Το άλλο σημαντικό που πρέπει να ακούσουμε είναι πως δεν πρέπει να πιστεύουμε όλα όσα ακούμε για τα ορυχεία της Κίνας. Αυτή είναι μια φωτογραφία ανθρακορυχείου που παράγει γύρω στους 15 εκατομμύρια τόνους το έτος βαθύ ορυχείο. Μιλάμε για πέντε φορές μεγαλύτερο από τα μεγαλύτερα ορυχεία της Ευρώπης. Ναι, υπάρχουν μικρά επικίνδυνα ορυχεία που θέλει να κλείσει η κινέζικη κυβέρνηση, αλλά αυτά τα μεγάλα ορυχεία αυξάνουν την παραγωγή και είναι πιο παραγωγικά από τα ορυχεία οπουδήποτε αλλού στον κόσμο και με προδιαγραφές ασφαλείας που είναι εξίσου υψηλές με τις δύσεις. Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Τα κυρία πλέον του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα επιμείνω γιατί είναι προφανή νομίζω. Είναι η βασική επιτόπια πηγή ενέργειας, εάν βεβαίως ε, δεν ε, υπολογίσουμε τις ΑΠΕ και την ενεργειακή αποδοτικότητα, μιλάμε για 80% των αποθεμάτων. Ο άνθρακας και ο λιγνίτης βρίσκονται σε πάρα πολλά κράτη-μέλη, στα περισσότερα θα έλεγα, αλλά μπορώ να πω και σε πολλά νομίζω. Φτάνει αυτό. Εξισορροπεί το ενεργειακό μείγμα της Ένωσης, λύνει ζητήματα ασφάλειας εφοδιασμού και τιμών. Και τα ορυχεία και όλη αυτή η αλυσίδα του πλούτου που δημιουργούν είναι πάρα πολύ σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά για μειονεκτικές περιοχές και απασχολούν γύρω στα 280.000 άτομα. Δεν θα καθίσω εδώ πέρα βεβαίω, ε, να δυσφημίσω άλλα καύσιμα, αλλά πρέπει να πω πω όλε οι πρωτογενείς πηγές ενέργειας έχουν τα υπέρ και τα κατά. Αυτά τα οποία έχω γράψει εδώ πέρα είναι τα πλεονεκτήματα του άνθρακα. Το βασικό μειονέκτημα είναι σαφές. Είναι οι εκπομπέ. Αλλά και άλλες πηγές ενέργειας έχουν τα μειονεκτήματά του. Θα εστιάσω λίγο στη Βουλγαρία. Θα μπορούσα να αναφερθώ και σε άλλα κρατημέλη. Ε, παρόμοιες καταστάσεις στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Αλλά αυτό το οποίο έχουμε εδώ πέρα είναι μία εικόνα του ορυχείου στο Μίνι Μαρίτσα Ιστοπ στη Βουλγαρία όπου παράγεται το 33% του ηλεκτρισμού της Βουλγαρίας. Ξεκίνησε η εξόριξη πριν από 50 χρόνια και τα σημερινά σχέδια εκτείνονται μέχρι το 2070. Μιλάμε για 60 χρόνια στο μέλλον. Η AES, η Αμερικανική εταιρεία ηλεκτρισμού, χτίζει ένα νέο σταθμό παραγωγής ενέργειας, ενώ άλλοι σταθμοί έχουν αναβαθμιστεί για να συμμορφωθούν με τις οδηγίες εκπομπών των οδηγιών της Ένωσης. Λίγα λόγια για το άλλο ερώτημα, εάν μπορεί να είναι καθαρός ο άνθρακας. Μπορούμε βεβαίω να αφιερώσουμε μια ολόκληρη ακρόαση σε αυτό το ζήτημα στη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Θα αναφέρω λίγα πράγματα μόνο. Βλέπετε μια φωτογραφία εδώ Μια σειρά εργοστασίων παραγωγής ενέργειας που είναι το ένα δίπλα στο άλλο στη Δανία. Σημαντικό είναι να πούμε πως τα νεότερα πιο αποτελεσματικά εργοστάσια έχουν μικρότερες εκπομπές αναμονάδα παραγόμενου ηλεκτρισμού, κάτι το οποίο πρέπει να ενθαρρύνουμε να αντικαταστήσουμε τα παλαιότερε τις παλαιότερες μονάδες με νεότερες. Βλέπετε εκεί πέρα μια γραμμή η οποία έχει μια τάση κατηφορική, δείχνει τις εκπομπές αναμονάδα ηλεκτρισμού. Βλέπετε, είναι υψηλός ο παγκόσμιος μεσόρος, λίγο καλύτερος ο ευρωπαϊκός μεσόρος, η τελευταία τεχνολογία λίγο πιο χαμηλή, η τελευταία τεχνολογία μπορεί να φτάσει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα και βλέπετε δέσμευση και αποθήκευση πόσο μεγαλύτερη βελτίωση εκπροσωπεί. Αλλά κάποια από τα καλύτερα εργοστάσια είναι στην Ευρώπη. Παραδείγματο χάρη η Δανία παράγει το μισό τη ηλεκτρισμό από άνθρακα σε πολύ αποτελεσματικά εργοστάσια. Αυτό το οποίο είναι στα δεξιά εδώ πέρα είναι πιθανώ το αποτελεσματικότερο στον κόσμο μια αποτελεσματικότητα του 47%. Η Ιαπωνία, Κορέα και άλλες ασιατικέ χώρες έχουν κάποιε από τις πιο σύγχρονες και καθαρότερες μονάδες. Δεν θα μιλήσουμε σε βάθος για τη δέσμευση και αποδίκευση, αλλά εξυπακούεται πω εν ευθέτω χρόνο το διοξείδιο του άνθρακα θα πρέπει να δεσμεύεται και να αποθηκεύεται υπογείω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει εδώ πέρα ηγετικό ρόλο και αυτό το καλωσορίζει ο κλάδος μας ε, και η βιομηχανία μετάδοσης ηλεκτρισμού και πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις. Οπότε θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε τις μονάδες παραγωγής και να έχουμε νέα εργοστάσια τα οποία θα δεσμεύουν και θα αποθηκεύουν κατευθείαν. Οπότε, για να απαντήσω στα ερωτήματα που έθεσα. Εάν είναι ο άνθρακα καύσιμο του μέλλοντος, ναι, είναι η πηγή ενέργεια η οποία αναπτύσσεται ταχύτερα στον κόσμο. Ανεξαρτήτως του τι θα κάνει η Ευρώπη, ο άνθρακα είναι καύσιμο του μέλλοντος στον κόσμο. Δεύτερον, μπορεί να είναι καθαρό, ναι, είναι ασφαλή, αξιοπιστο, φθηνό, γίνεται όλο και πιο αηφόρο και μπορούμε να επιτύχουμε χαμηλέ εκπομπές με δεσμευτική αποθήκευση. Χρειάζεται η Ευρώπη τον άνθρακα, ναι, μας δίνει τη δυνατότητα ποικιλία είναι επιτόπιο καύσιμο, μειώνει την ενεργειακή εξάρτηση και δημιουργεί πλούτο. Οπότε για να επιτύχουμε τις προκλήσεις που έχουμε θέσει θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πολλές τεχνολογίες. Πυρηνική, ανανεώσιμες, δέσμευση και αποθήκευση και στο φυσικό αέριο και στον άνθρακα και χάρηκα για το ότι χτες στο Ηνωμένο Βασίλειο η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως και το φυσικό αέριο θα αποτελέσει κομμάτι του ε, ε, έργου επίδειξης δέσμευσης και αποθήκευσης. Οπότε ο άνθρακα αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του ενεργειακού μείγματο και η Ευρώπη έχει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τα αποθέματα άνθρακα και λιγνίτη με τρόπο που θα αποτελέσει υπόδειγμα για όλο τον πλανήτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίε και κύριοι. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τον λόγο τέλος και έχουμε ένα πρόβλημα λίγο χρόνου τον κύριο Τζόνσον από την βέβαια την Μονάδα Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Let's Σε ελπίσουμε ότι θα λειτουργήσει το μηχάνημα. Um, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας μιλήσω. Προχωρώ και δεν ξέρω αν ε, το βλέπετε εκεί στο τέλος. Στο τέλος του τίτλου της ομιλίας μου προσέθεσα και ένα ερωτηματικό. Ο ρόλος του άνθρακα στο μελλοντικό ενεργειακό μείγμα. Ερωτηματικό για μας είναι ερωτηματικό. Δεν είμαστε κατά ανάγκη κατά του άνθρακα ή των ορυκτών καυσίμων, αλλά ο ρόλος του άνθρακα, μακροπρόθεσμα, αν έχει μακροπρόθεσμο μέλλον, θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα και αν είναι δυνατόν, αν θα μπορέσει να αποκριθεί με τη μόλυνση. Χωρίς να αγνοούμε την κοινωνική, οικονομική σημασία του άνθρακα, τόσο στο παρόν όσο και στο παρελθόν, κυρίως στην Ευρώπη και σε άλλες πλούσιες περιοχές του κόσμου, θεωρούμε ότι τελικά το μέλλον του θα εξαρτηθεί από την επιταγή της προστασίας ε, του ε, κλίματος από περαιτέρω ζημιά. Μιλάμε για μια ακρόαση περί του άνθρακα, όχι για το κλίμα. θα μιλήσω για τη, τα θέματα σε σχέση με το κλίμα και μετά θα μιλήσω για τον άνθρακα. Θα μπορούσα να σας δείξω πολλά σχεδιαγράμματα, αλλά ήδη έχετε δει πολλά. Σε σχέση με την κλιματική αλλαγή όμως, ποια είναι η κατάσταση που εμείς ή και ολόκληρος ο κόσμος έχει να αντιμετωπίσει. Ο καλύτερος τρόπος να το απεικονίσω αυτό εδώ στις Βρυξέλλες είναι αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρος Μπαρόζο στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Επιχειρήσεων πριν από περίπου ένα χρόνο, υπάρχει στη διαφάνεια. Η κλιματική αλλαγή είναι το υπαριθμόν ένα καθοριστικό θέμα της γενιάς μας. Είναι το υπαριθμόν ένα και το πιο η πιο υπαρξιακή ε, πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Η πιο υπαρξιακή πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, είπε ο πρόεδρος Μπαρόζο. Χωρίς να μπούμε σε νούμερα, αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Όχι μόνο σε σχέση με την τροχιά που θα ακολουθήσουν ε, το της ενέργειας τα επόμενα 50 χρόνια, αλλά και ολόκληρη η οικονομία και ολόκληρες οι κοινωνίες μας, αν δεν λύσουμε το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής οι, δυνα... το... δυνατότητες καταστροφής και βλέπουμε τα φαινόμενα σε ολόκληρο τον κόσμο αυξάνονται αν δεν αντιμετωπίσουμε την επιταγή της... Ε, που μας επιβάλλει η κλιματική αλλαγή. Το κλιματικό ζήτημα δεν είναι βεβαίω τόσο επίκαιρο τώρα όσο πριν από ένα χρόνο. Και όλοι γνωρίζουμε τον λόγο. Βρισκόμαστε στα πλαίσια μιας ε, διεθνούς ε, πολιτικής διαδικασίας και ως εκ τούτου δεν είναι τόσο επίκαιρο, αλλά η κατάσταση, όσον αφορά την κατάσταση της ατμόσφαιρας, οι προστίκες στην ατμόσφαιρα και αυτό που λένε οι ειδικοί επιστήμονες για την τάση που εμφανίζεται στην ατμόσφαιρα. Αυτά τα θεμελιώδη ζητήματα δεν εξαφανίστηκαν, ας μην παρόλο που δεν τα συζητάμε και τόσο πολύ πια. Στα γρήγορα λοιπόν, ποια είναι η ε, γενικές οριακές καταστάσεις για το, για το μέλλον της οικονομίας. Περιορισμό ε, περιορισμός κατά 1,5% μόνο της υπερθέρμανσης πάνω από το μέσο όρο. Τι σημαίνει αυτό όσον αφορά τις εκπομπές προς την ατμόσφαιρα. Σημαίνει ότι μέχρι, από τώρα μέχρι τα μέσα του αιώνα περίπου όλος ο κόσμος για να αποφύγει η επικίνδυνη κλιματική αλλαγή έχουμε μόνο ένα τρισεκατομμύριο ε, ε, αντίστοιχα εκπομπών που πρέπει να εκπαιμφθούν. Αλλά επίσης, εκτός από τους στόχους, πρέπει να μιλήσουμε και για τις συγκεντρώσεις εκπομπών και όσον αφορά τους στόχους της δικής μας περιοχής, πρέπει να δούμε πώς ε, εντάσσονται, πώς ταιριάζουν ένας με τον άλλον. Στην Ευρώπη λοιπόν γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα μακροπρόθεσμο στόχο για το πού προχωρούμε, προς τα πού πηγαίνουμε. Πέρυσι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενώψη της Κοπενχάγης δεσμεύτηκε στο 80 95% μείωση των εκπομπών για την Ευρώπη μέσα σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο όπου παρόμοιες οικονομίες θα κινηθούν ανάλογα. Επίσης, ταυτόχρονα περίπου Πέρυσι είχαμε την δέσμευση του Πρόεδρου Μπαρόζο στις κατευθυντήριες γραμμές του κατά την παρουσίαση της δεύτερης θητείας του και συζητήθηκε, συζήτησε στο Κοινοβούλιο όταν ενέκρινε το Κοινοβούλιο τη δεύτερη θητεία του ότι η Επιτροπή Μπαρόζο 2 θα κάνει τα πρώτα βήματα για να απανθρακώσει, να αφαιρέσει τον άνθρακα μάλλον από τον τομέα της ενέργειας, να αφαιρέσει πλήρως τον άνθρακα από τον τομέα της ενέργειας. Και βεβαίως ε, η Κομισιόν όπως ε, γνωρίζετε η Κομισιόν δουλεύει για έναν ε, οδικό χάρτη για το 2050 για την ενέργεια που θα αρχίσει να τον παρουσιάσει στις αρχές του επόμενου έτους και να τον αναπτύσσει στη διάρκεια του έτους. Τώρα αυτά μήπως είναι λόγια απλώς, πολιτικές εξαγγελίες. Θέλω να σας δείξω πώς οι υψηλού στόχοι διαμορφώνονται σε σχέση με την πολιτική που αναπτύσσεται αρκετά κοντά ε, στο ξενοδοχείο που βρίσκεται εδώ απέναντι. Την άνοιξη φέτος ο Φίλιπ Λόου, γενικό ο διευθυντής της Γενικής Ενέργειας, αναφερόμενος ε, μιλώντας στην ετήσια συνάντηση της ε, βιομηχανίας άνθρακο, είπε ότι η αφαίρεση του άνθρακα είναι εξαιρετική σημασία και ότι το CCS είναι απαραίτητο για την επιβίωση του άνθρακα. Και τα δύο αυτά πρέπει να τα επαναλάβουμε αφαίρεση του άνθρακα είναι εξαιρετικά μεγάλη σημασία, είπε ο Γενικό Διευθυντή Ενέργεια, υπεύθυνο την ενέργεια και το CCS είναι απαραίτητο για την επιβίωση του άνθρακα. Σκεφτείτε το αυτό σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν με την προηγούμενη ε, διαφάνεια. Μιλάμε για πλήρη αφαίρεση του άνθρακα. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε λεπτομερέστερα, τι θα γίνει πότε, το, μέχρι το 2020, το 30 κλπ. Αλλά τελικά μιλάμε για πλήρη αφαίρεση του άνθρακα, αν πρόκειται να επιβιώσει ο άνθρακας στο πλαίσιο του ενεργειακού μείγματος. Εξ όσων, γνωρίζουμε η στρατηγική 2020 που, θα, που εγκρίθηκε από τους επιτρόπους σήμερα αν δεν κάνω λάθος και θα παρουσιαστεί αύριο δεν αναφέρει ρητά τον άνθρακα καθόλου. Όπως είπα στην αρχή της ομιλίας μου, εμείς δεν ε, αγνοούμε την κοινωνική και οικονομική σημασία του άνθρακα στο παρόν ενεργειακό μείγμα, αλλά σε σχέση με αυτό που λέει η Κομισιόν για την μελλοντική της στρατηγική, ο άνθρακας δεν αναφέρεται στο έγγραφο της Κομισιόν, αυτό που θα παρουσιαστεί αύριο το πρωί. Πιο συγκεκριμένα για τον άνθρακα τώρα. Καταρχήν δεν είμαστε κατά τη χρήση των ε, ορυκτών καυσίμων. Αλλά μας απασχολεί ότι δεν υπάρχει ισότητα μεταχείρισης. Φέτος έγινε μια συζήτηση μεταξύ των θεσμικών οργάνων, ψηφίστηκε σήμερα το πρωί εδώ, ε, μια προθεσμία για να ε, λήξουν οι εθνικές λειτουργικές επιδοτήσεις η ύπαρξη αυτών των ε, επιδοτήσεων στην Ευρώπη δεν είναι ισοδύναμη. Μερικές χώρες, μεταξύ των οποίων η Τσεχία, η Πολωνία, ε, έχουν ε, ανταγωνιστική παραγωγή άνθρακα, άλλες όχι. Αυτές οι επιδοτήσεις πρέπει σύντομα να σταματήσουν. Τα θεσμικά όργανα και κυρίως το Συμβουλίο Υπουργών και η Κομισιόν, όπως υπογράμμισαν, συμφωνώ μαζί σας και το είπα πριν σε άλλες χώρες όμως δεν ισχύει αυτό που λέτε. Τα θεσμικά όργανα θα θέσουν προθεσμία για να λήξουν αυτές οι λειτουργικές ενισχύσεις. Οπότε πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτούμε τους άλλους τρόπους με τους οποίους η μόλυνση και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του άνθρακα θα περιοριστούν. Το σύστημα ETS υπάρχει, αναθεωρήθηκε η οδηγία ETS πριν από δύο χρόνια. Εξακολουθούμε όμως να βλέπουμε ότι το ETS είναι ένα εργαλείο πολιτικής που εξακολουθεί να είναι αδύναμο και δεν μπορεί να περιορίσει τις εκπομπές άνθρακα και άλλων ορυκτών καυσίμων στο πλαίσιο αυτών των οριακών ε, προϋποθέσεων για την κλιματική αλλαγή. Δεν ε, πρέπει να το καταργήσουμε ή να το αλλοιώσουμε, το ETS, αλλά πρέπει να το κάνουμε αποτελεσματικό το μέσο αυτό. αυτό είναι ένα από τα θέματα που μας απασχολούν. Το ανώτατο όριο πρέπει να μειωθεί. Θα βοηθούσε όλους όσοι ασχολούνται με την θέσπιση πολιτικής και τους βιομηχανικούς παράγοντες στον τομέα της ενέργειας να γνωρίσουν ότι το ETS είναι ένα ανοιχτό εργαλείο. Το δίκαιο του ETS δεν αναφέρεται στην τρίτη φάση, παρότι συχνά τη συζητάμε, τη λεγόμενη τρίτη φάση. Ο νόμος, χωρίς την παραμικρή αλλαγή, θα μειώσει το ανώτατο όριο κάθε χρόνο και θα φτάσει στο 0 περίπου το 2070 σε σχέση με τη γενική κατάσταση του κλίματος αυτό δεν είναι γρήγορα, δεν είναι αρκετά εγκαίρος. Πρέπει να συμβεί πριν από το 2050 και αυτή είναι μία από τις μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες. Επίσης για το ETS πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα αντισταθμιστικά ε, έγγραφα είναι ειλικρινή, είναι αυθεντικά και ότι περιμένουμε από την Κομισιόν ε, γρήγορα προτάσεις για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα της ε, ποιότητας και την ε, αυθεντικότητα των εγγράφων αυτών στην, στην Ινδία. Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις αράζουν, αλλάζουν τα μοντέλα παραγωγής για να επωφεληθούν από το αντισταθμιστικό όφελος που παράγεται εδώ κυρίως στην Ευρώπη αυτό είναι σκάνδαλο που πρέπει σύντομα να αντιμετωπιστεί και πρέπει η Κομισιόν γρήγορα να υποβάλει προτάσεις να στηριχθούν τα κράτη-μέλη σε αυτό το χώρο. Επιπλέον, σε αυτή τη διαφάνεια δεν ανέφερα ότι το CCS ε, το δέχεται η ΒΒΕΦ, αλλά στο πλαίσιο ενός αποτελεσματικού ε, νομιθωτικού πλαισίου όπου να πραγματοποιούνται οι ε, επιχειρήσεις του CCS το πακέτο που θεσπίστηκε προδιετίας είναι καλό, συνδέεται με άλλα κομμάτια περιβαλλοντικής νομοθεσίας και όσο τηρείται το CCS είναι αποδεκτό από εμά. Επανέρχομαι στις επιδοτήσεις του άνθρακα για λίγο. Είναι πολιτικό ζήτημα ποια θα είναι η ημερομηνία που θα μας πούν στο τέλος, ίσως αυτό οριστεί στη διάσκεψη κορυφής και όχι ε, σε επίπεδο Υπουργών Ανταγωνιστικότητας, το Δεκέμβρη δηλαδή. Η ΒΒΕΦ σαφώς ζητά από τα, κράτη, από τα μέλη του Κοινοβουλίου και τα άλλα θεσμικά όργανα που τυχόν παρίστανται να στηρίξουν την πρόταση της Κομισιόν χωρίς βασικές αλλαγές. Οι ενισχύσει λήγουν το 2014. Οποιαδήποτε παράταση δεν ε, μας βρίσκει, δεν βρίσκει σύμφωνα τα άλλα θεσμικά όργανα. Κυρίως η ημερομηνία του 2018 που προέκυψε από τη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων θα πρέπει να απορριφθεί στην Ολομέλεια. Ακόμα πιο ενδιαφέρον και αντιλαμβάνομαι ότι μου μένουν ελάχιστα λεπτά. Αν ε, σταματήσουμε τις άμεσες επιδοτήσεις, δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε νέες επιδοτήσεις, οι οποίες θα καταβάλλονται έμεσα. Πράγμα που έτσι ε, προτείνεται να γίνει αυτή τη στιγμή στην Ισπανία. Οι δύο κύριοι που βρίσκονται στην εικόνα αυτή, ο Μπαρόζο και ο Αλμούνια προώθησαν την Επιτροπή Οικολογίας το Σεπτέμβρη με λίγη υποστήριξη από τους συναδέλφους τους, χωρίς αντίρρηση από την Ισπανική κυβέρνηση, ένα μέρος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ισπανία να παραμείνει σε, με αποκλειστική χρήση του εσωτερικού παραγόμενο άνθρακα. Αυτή η απόφαση ανακλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την προηγούμενη εβδομάδα εν ώψη μιας ακρόασης για την νομιμότητα της απόφασης της Κομισιόν που βεβαίως θέτει υπό αμφισβήτηση την νομιμότητα της ισπανικής πρότασης. Εάν, και εδώ ε, φτάσαμε στην τελευταία μου διαφάνεια, αν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποια από τα θέματα που ανέφερα, την ε, μεταρρύθμιση του EPS, το τέλος, να λήξουν οι εθνικές επιδοτήσεις, να μην υπάρξουν ε, άλλες επιδοτήσεις που θα μπουν ε, την πίσω πόρτα και τη δυνατότητα για τις περιβαλλοντικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις να προκαταλάβουν κάποιες εξελίξεις, τότε το μολυντικό πλαίσιο του άνθρακα υπάρχει. Όπως σας είπα, το ΒΒΕΦ συμφωνεί με το CCS υπό την προϋπόθεση ότι η κυριαρχούσα ανάγκη για να ληφθεί υπόψη το κλίμα θα ε, στηριχθεί. Είμαστε ρεαλιστές, όχι δογματικοί και ίσως τα ETS θα είναι αποτελεσματικά ώστε να αναπτυχθεί επαρκώς η τεχνολογία CCS, ε, της δέσμευσης και αποθήκευσης δηλαδή. Η συζήτηση για την οδηγία έκλεισε το καλοκαίρι, αλλά αν, θα, αν ξανανοίξει στο μέλλον θα πρέπει ίσως να συζητήσουμε μια κανονιστική, κανονιστική νομοθεσία όπως έχουμε για τα νητρικ, τους νητρικούς ρήπους έτσι ώστε το καθαρός άνθρακας να φύγει από το σύστημα και κατά τον ίδιο τρόπο και άλλοι ρήπη. Αν οι ενεργειακές επιχειρήσεις, οι εταιρείες θέλουν να χρησιμοποιούν τα ε, ορυκτά καύσιμα με CCS, να υπάρχει, με CCS, υπάρχει τρόπος συγκεκριμένος που να μπορούν να το κάνουν αυτό. Ενώ το ETS, αυτό ίσως είναι πολύ σύνθετο που θέλω να σας πω, πολύ μπερδεμένο και ίσως να μην το ξεκινήσω. Εν πάση περιπτώσει, όσο παραμένουν ανώριμα τα ETS και όσο δεν υπάρχει επαρκής ανταπόκριση στα θέματα του κλίματος, είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που τους δίνουν η, τους δίνει το κεφάλαιο 3 της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια που τη γνωρίζετε με βέβαιος για αυτές οι εξουσίες σε επίπεδο ε, κράτους μέλους για τη συγκατάθεση σε νέα, για νέα δυναμικότητα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με σοφροσύνη ώστε να αποφύγουμε τη δημιουργία νέων σταθμών παραγωγής που να έχουν υψηλές εκπομπές σε άνθρακα. Δηλαδή να μην βρεθούμε στο μέλλον σε μια κατάσταση που θα έχουμε μεγαλύτερη δυσκολία να ανταποκριθούμε στις επιταγές της κλιματικής αλλαγής επειδή σήμερα πήραμε λάθος αποφάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ομιλητές. Τελειώσαμε με τις συνεισφορά σας. Θα ακούσουμε κάποιες ερωτήσεις και μετά θα τοποθετηθεί και η Κομισιόν. Έχουμε δέκα λοιπόν συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο. Δύο λεπτά ο καθένας παρακαλώ. Αλλιώ δεν θα τα καταφέρουμε. Κύριε Καρβάγιο, λοιπόν, πρώτα. I would like to thank all the... Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου του ομιλητέ. Πολλοί μίλησαν πάρα πολύ για την αποδοτικότητα και το διοξείδιο του ανθρακά, για την ποιότητα του αέρα. Υποθέσατε ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Ξέρω πως έχει γίνει πάρα πολύ έρευνα, αλλά περισσότερες από τις υπάρχουσες τεχνολογίες είναι άκριβες και στις περισσότερες χώρες δεν χρησιμοποιούνται οι υπάρχουσες ε, τεχνολογίες. Και γεγονός είναι πως για το μονοξίδιο του αζότου, για τα οξύδια του αζότου, πάρα πολλά έχουν γίνει, επανακάψη κτλ. Αλλά για τα αιρούμενα σωματίδια και τα βαρέα μέταλλα υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Και αναρωτιέμαι ποιες είναι οι λύσεις και ποια είναι η άποψή σας. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνα για την υγεία. Δεύτερο ερώτημα για τα πολύ κρίσιμα έργα τα οποία τρέχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό το, το έργο αυτό. Ήμουν ερευνήτρα εγώ και είχα εργαστεί εγώ στην Γενική Διεύθυνση 17 πάνω σε αυτό το θέμα. Πώς θα προχωρήσει πιο γρήγορα το έργο. Ποιο είναι το πρόβλημα, τα υλικά και η θερμοκρασία. Τελευταίο ερώτημα. Εξετάσαμε πρόσφατα την διαθεσιμότητα του άνθρακα. Την προηγούμενη εβδομάδα η Νότιος Αφρική έβγαλε μια έκθεση που λέει πως ε, τα αποθέματα που νόμιζαν ότι είχαν είναι χαμηλότερα από όσο νόμιζαν. Αυτό είναι μόνο νοτιοαφρικανικό. Νοτιοαφρικανικό ζήτημα Εγνωρίζετε και άλλα τέτοια ζητήματα για διαθεσιμότητα του άνθρακα. Τέλος, για τον κύριο Τζόνσον, συμφωνώ για τις ανησυχίες που έχετε για τα βιομηχανικά αέρια. Χτες ζήτησα από τον Επίτροπο, την Επίτροπο για το κλίμα τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει, όχι μόνο για το μάλλον μέσω του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης, αλλά άμεσα να μην ε, αναγκαστούμε να έχουμε όλες αυτές τις άδειε προκύπτουν από την Κίνα. Και η Επίτροπος ήταν πάρα πολύ θετική, είπε πως οι υπηρεσίες της το μελετάνε. Για να δουν πώς θα λύσουμε το πρόβλημα, για να μην είμαστε αναγκασμένοι να αποδεχτούμε όλες αυτές τις ε, άδειε που τι θα κάνουν ουσιαστικά να μεταφέρουν χρήματα από την Ευρώπη στην Κίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι σύντομος. Δεν συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τζόνστον για το θέμα δέσμευσης και αποθήκευσης. Η έκθεση Davis πρέπει να αλλάξει. Είναι ανεπαρκής, ακατάλληλη, γιατί αποκλείει την κατασκευή πιο αποτελεσματικών μονάδων, αποτελεσματικών κατά 60-70%. Η δέσμευση και αποθήκευση θα εισαχθεί για διάφορα καύσιμα. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Μήπως θα ήταν καλό να έχουμε νομοθεσία η οποία θα επιτρέπει την οικοδόμηση νέων σταθμών με βαθμό αποτελεσματικότητας πάνω από 50% ανεξαρτήτως της κατάστασης με τη δέσμευση και αποθήκευση γιατί ο Ντέιβις υποθέτει πως οι σταθμοί με άνθρακα θα πρέπει να έχουν δέσμευση και αποθήκευση αλλιώς δεν μπορούν να φτιαχτούν. Ευχαριστώ η κυρία Ριέρα Μαδουρέλη. Ε, ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη, δεν σα άκουσα καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του ομιλητέ, σα άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον Το θέμα αυτό βεβαίω ε, έχει απασχολήσει πολλές φορές την Επιτροπή μας και την ομάδα μας. Το κλείσιμο τώρα των μη ανταγωνιστικών ανθρακοριχείων θεωρούν κάποιοι συνάδελφοι πως θα πρέπει να επιβραδυνθεί. Γνωρίζω όμως πάρα πολύ καλά τις οικονομικές συνέπειες σε κάποιες ε, περιοχές της Ένωσης εκεί όπου τα ανθρακοριχεία προσφέρουν και είναι βασική πηγή απασχόλησης, αντιλαμβάνομαι τους περιβαλλοντικούς ε, λόγους και τους λόγους ανταγωνιστικότητας που θέτουν κάποιοι συνάδελφοι ε, για να κλείσουν αυτά τα ορυχεία, αλλά για μένα είναι απολύτως απαραίτητο να σκεφτούμε τις δουλειές που θα χαθούν, τις θέσεις εργασίας, που θα χαθούν άμεσα. Εάν περιοχές αυτές δεν μπορέσουν να προσαρμοστούν. Πρέπει να δούμε τις θέσεις εργασίες που θα χαθούν. Και μετά από αυτά τα οποία μας είπατε, θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο εκμετάλλευση του άνθρακα για να γίνει λιγότερο ρηπογόνος και πιο ανταγωνιστικός. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Πρέπει να τονίσω τις προσπάθειες που έκαναν πολλές περιφέρειες να κλείσουν ορυχεία. Θα μπορούσατε ίσως να μας πείτε κάποια πράγματα περισσότερο για το τι ελπίδα μπορείτε να δώσετε σε αυτές τις ε, περιοχές. Μιλήσαμε για τα τα των ορυχείων, ε, ίσως να μην συμφωνούμε 100% ε, με τους συναδέλφους από την Πολωνία. Εσείς ε, μας είπατε την άποψή σας, το κόστος του πετρελαίου και τους μισθούς και τα λοιπά, θα μπορούσατε ίσως να μου πείτε τι ακριβώς θεωρείτε ένα ανταγωνιστικό ρηχείο. Και ε, είμαι υπεύθυνη επίσης για την έρευνα στην Επιτροπή, είμαστε εδώ πέρα και υποστηρίζω πάντα οποιοδήποτε έργο σχετίζεται με μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και βεβαίως ε, τον ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι λοιπόν βιώσιμο και αποδεκτό ε, βραχυπρόθεσμα Έχω και άλλες ερωτήσεις ε, και θα ήθελα να συνεχίσω, αλλά έχει τελειώσει ο χρόνος. Με ευχαριστώ, κυρία Βάγκνερ. Primero felicitar a los cuatro ponentes porque han sido muy Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, ε, παρεμβαίνοντες. Πολύ ενδιαφέρον αυτό αυτά που μας είπε πολύ σύντομες ερωτήσεις. Αν μπορούν να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες και περισσότερες αποσαφηνήσεις όσον αφορά την ε, έρευνα, ε, ε, όσον αφορά την δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και την, την δυνατότητα δημιουργίας εγκαταστάσεων για το σκοπό αυτό, καθώς επίσης και μια ιδέα κόστους, οικονομικού κόστους. Δεύτερον, αν υπάρχουν ε, διαφορές ποιότητας ε, στους ε, διάφορους τύπους άνθρακα που έχουμε στην Ευρώπη. Ο κύριος Πόλα που προέρχεται από μια περιοχή που αγαπάω πάρα πολύ θα μπορούσε να μας πει κάτι. Κύριε Στούρμα, ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση στον κύριο Πίκατς. Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα, ε, σας ευχαριστούμε που είσαστε υπέρ της ε, βελτίωσης του κλίματος, γιατί δεν είναι όλοι όσοι εκπροσωπούν ε, την ανθρακοβιομηχανία. Μας λέτε ότι θα βελτιωθεί η τεχνολογία έτσι ώστε το, ο άνθρακας να έχει μέλλον. Αλλά τον Οκτώβριο το τελευταίο σενάριο ας πούμε που έκανε η Κομισιόν λέει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ε, κάποιο πρόγραμμα που να λέει ότι ότι εάν φτάσουμε σε ένα επίπεδο δέσμευσης αποθήκευσης άνθρακα του 20% ε, και αν χρησιμοποιήσουμε και ανανεώσουμε πηγές ενέργειας, ότι θα μπορέσουμε ε, να ε, βελτιώσουμε τα αποτελέσματα στο μέλλον. Και εξάλλου είναι κάτι που κοστίζει πάρα πολύ. Εσείς είστε κατά του να πάμε από το 20% στο 35% γιατί ενδεχομένως θα αυξηθούν οι τιμές του άνθρακα. Τώρα, εάν ε, δημιουργούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις μέσω ε, συμβάσεων ε, στην αγορά, τότε θα δημιουργείται μια αγορά για την δέσμευση και την αποθήκευση του άνθρακα και ε, τότε θα μπορούσαμε ε, να ε, βάλουμε τον όρο της αποθήκευσης για οποιαδήποτε επένδυση και τότε θα ήταν λογικό να μπαίνουν οι όροι αυτοί, θα υπήρχε δηλαδή ένα μέλλον για αυτούς τους στόχους. Υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει Υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνω. Εάν ε, δεν μας βοηθήσετε να ε, ε, δεχόμενοι κάποιες υποχωρήσεις αρχικές, έτσι ώστε πραγματικά να υπάρχει ανάγκη επιχειρηματική για δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα, τότε δεν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε αυτή την στρατηγική για το CCS. Εσείς προτείνετε να έχουμε τεχνολογική λύση. Και λέτε ότι θα πρέπει να ε, συνεχίσει η διαδικασία, να γίνουν δηλαδή πιο πράσινες οι εκπομπές ε, από τις ε, εγκαταστάσεις, από τις μονάδες παραγωγής που χρησιμοποιούν τον άνθρακα. Αλλά να σας πω, εάν η Γερμανία εάν το 95% ε, του στόχου αυτού της μείωσης της Γερμανίας. Εάν πετύχει 50 με 60% ε, των εκπομπών ε, θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι το 15. Τότε εσείς ανοίγετε την πόρτα για την συνέχιση δημιουργίας Ε, να συνεχίσει η παραγωγή μέσα από παραδοσιακές μονάδες. Κρίστιαν Ήλα, επόμενη ερώτηση. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για το ότι δεν μας λέτε αυτά τα οποία λέει συνέχεια ο Τούρμες, αυτή η εθνοκεντρική άποψη του κόσμου. Συνέχεια εθνοκεντρικά στην Ευρώπη και αγνοεί πλήρως τις διεθνείς εξελίξεις. Πριν από 14 ημέρες η Κίνα δημοσιοποίησε ένα στρατηγικό σχέδιο για να αποκτήσει πλειοψηφικά πακέτα σε διεθνή ανθρακοριχία. Ο δε κύριος Μετβέντεφ πριν από τρεις μήνες είπε πως η Ρωσία στις προοπτικές μελλοντικέ για την συνολική παραγωγή ρεύματο θέλει να μεταβεί σε μονάδες άνθρακα και να γίνει μάλιστα και εισαγωγέα άνθρακα. Οπότε είμαι πεπισμένος πως εάν είναι να πετύχουμε κανένα κλιματικό στόχο σε διεθνές πλαίσιο και να μην οδηγηθούμε απλά σε οικονομική καταστροφή της Ευρώπης, που θα είναι και οικολογική καταστροφή ταυτόχρονα, θα πρέπει να τεθεί το ερώτημα των αποτελεσματικών ε, εργοστασίων άνθρακα και της ε, δέσμευσης. Δύο ερωτήματα. Πρώτον, είναι ενδιαφέρον από πλευρά οικονομική το ποια είναι η εξέλιξη της τιμή του άνθρακα με βάση αυτά τα οποία σας είπα. Ποιε είναι οι εκτιμήσει σας δηλαδή. Είπατε ο άνθρακας είναι μια φτηνή τεχνολογία κτλ. Αλλά ισχύει αυτό δεδομένου π.χ. δεδομένης της στενοπού που αντιμετωπίζουμε στην παροχή αερίου παραδείγματο χάρη εμεί στην Ευρώπη. Το πρώτο ερώτημα αυτό. Δεύτερο ερώτημα και δεν είναι τελείω λάθος αυτό το οποίο Κλοντ Τούρμες. Πώς εκτιμάτε αυτή τη στιγμή το θέμα της εξέλιξης τη τιμή στο πλαίσιο της δέσμευσης και αποδίκευση κομισιών το, τοποθετήθηκε το εάν είναι σωστό είναι ένα άλλο ερώτημα αλλά θα ήθελα να ακούσω τη δική σας απάντηση και τρίτο ερώτημα πόσο μεγάλη θεωρείται την πιθανότητα στην Ευρώπη, στα κράτη-μέλη, να υπάρξει εφαρμογή ε, οδηγιών δέσμευσης και αποδικευσής, γιατί διαφέρει πάρα πολύ η ε, κατάσταση και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τις επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα. Ωραία. Τώρα έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να απαντηθούν αυτές οι ερωτήσεις. Προτείνω να πάμε με τη σειρά. ξεκινήσουμε με τον κύριο Τζόνσον, ο οποίος μίλησε τελευταίος και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να προσπαθήσετε ε, να απαντήσει ο καθένας κάποιες ερωτήσεις και να επικεντρωθείτε σε αυτές. Κύριε Τζόνσον. Um, μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης, όπως είπατε, συμφωνούμε. Υπάρχουν δύο επίπεδα στα οποία ρυθμίζεται αυτή η αγορά. Το ένα είναι το παγκόσμιο και το άλλο είναι το ευρωπαϊκό. Και δεν υπάρχει συμφωνία στο παγκόσμιο επίπεδο. Μπορούμε όμως να επιδείχουμε συμφωνία στο ευρωπαϊκό επίπεδο που υπάρχει ήδη κάποιο αποθεματικό στην οδηγία και κάποιες εξουσίες που επιτρέπουν στην Κομισιόν να το κάνει. Επί νομίζω συμφωνούμε. Είναι θέμα των κατάλληλων μονάδων να κινηθούν. Ο κύριος Γκέρεκ δεν είναι εδώ. Να απαντήσω όμως για τα πρακτικά, εν περιπτώσει. Νομίζω πως συμφωνούμε ε, στην ερμηνεία της οδηγίας γεωλογικής αποθήκευσης μέρος οποίας απαιτέρεσε η έκθεση Chris Davis. Εάν είναι εδώ βοηθός του ή αν θέλει να δώσει κάποια συνέχεια, μπορώ να το κάνω αυτό. Πρόσωπο με πρόσωπο για να δούμε το τι λέει και τι δεν λέει η οδηγία. Η κυρία Ριέρα Μαδουρέλ, τι ελπίδα υπάρχει στην Ισπανία και ειδικά στις ε, περιοχές εκείνες της Ισπανίας που πλήττονται από την παρακμή αν θέλετε του Ανθακά έχω αντιληφθεί πως ε, στον τομέα της παραγωγής υπάρχουν 4.000 θέσεις εργασίας ο τομέας των ανανεώσιμων ο οποίος αναπτύσσεται γρήγορα όμως στην Ισπανία και έχει την πολιτική στήριξη της Ισπανίας και πρέπει να το πούμε αυτό αντιλαμβάνομαι πως εκεί πέρα υπάρχουν 200.000 θέσεις εργασίας στη χώρα σας στον τομέα αυτών Τότε η ενέργεια ένας τομέας ε, βιομηχανικός όπως η ενέργεια ποτέ δεν μένει στάσιμος και υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα ζητήματα βέβαια με την Ισπανία και τον Άνθρακα αυτή τη στιγμή όπως είπα η Ισπανία πρέπει να αναγνωρίσουν πως έχει επιτυχία στον τομέα των ανανεώσιμων και terms για την δέσμευση και αποθήκευση ειδικά είπα λέω συνήθως πως δεχόμαστε τη δέσμευση αποθήκευση. Δεν σημαίνει πως την στηρίζουμε, είναι κάτι το διαφορετικό. Το δέχομαι είναι κάτι παθητικό. Το στηρίζω είναι να την υποστηρίξουμε με, σε διάφορα φόρα. Η αποδοχή είναι κάτι διαφορετικό. E για το EPS και για άλλα ζητήματα αριθμιστικά ναι, αφέρθηκα σε αυτό γιατί τελείωσε ο χρόνος, αλλά ήταν στις διαφάνειες. Θα το ξέρετε βεβαίω γιατί ήταν και ο σκιώδης ηγητής στην οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές. Ιδεοδό θα έπρεπε να έχουμε τέτοιες προδιαγραφές ε, απόδοσης, ε, εκπομπών, κατά το οποίο συμφωνήθηκε χτες ατύπως στο Συμβούλιο για μια σειρά πολιτικών λόγων. Αυτή η νομοθεσία δεν είναι τόσο ισχυρή όσο θα μπορούσε να είναι, αλλά όπως σας είπα αναφέρθηκα στην ευκαιρία να ξανανοίξει κάτι τέτοιο στο μέλλον για να χρησιμοποιηθεί και για τον έλεγχο του κλίματος, όπως και για τον έλεγχο άλλων ακομπών. Και όσον αφορά την ανάσταση, εάν θέλετε, της ε, ευρωπαϊκής αυτής ε, πολιτικής διαδικασίας προστασίας του κλίματος, ναι, και αυτό θα πήγαινε εκεί πέρα. Αλλά πράγματι θα πρέπει να τονιστεί αυτό σε όλα τα ευρωπαϊκά, στα πολιτικά επίπεδα, σε αυτό συμφωνούμε. Και σε, θα μείνω σε αυτά. Ε, Ευχαριστώ, Πούλα Αλόνζο. Sí, muchas gracias, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Απαντώντας σε κάποιες από τις ε, ερωτήσεις και σε αυτές που απευθύνθηκαν σε μένα. Ε, όπως ε, σας έλεγα και προηγουμένως, τα τελευταία χρόνια οι μονάδες παραγωγής στην Ισπανία έχουν κάνει πάρα πολλές επενδύσεις ε, όσον αφορά την ε, δέσμευση και ε, αποθήκευση, όσον αφορά την αποθείωση. Έχουμε κάνει πάρα πολλές επενδύσεις και όταν έλεγα ε, για, όταν αναφερόμουν σε ενεργειακή ανεξαρτησία ε, αναφερόμουν σε ανεξαρτησία η οποία θα βασίζεται σε, σε σωστό, με σωστό τρόπο και επίσης ότι ε, διατείνομαι και πραγματικά το πιστεύω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να μην ε, εξαρτάται από τις μετατροπές της τις διακυμάνσεις της τιμής. Ε, στον ε, τομέα των, ε, της εξόρυξης έχουμε περάσει από 12 εκατομμύρια σε 1 εκατομμύριο τόνους. Έχουν μειωθεί στο μισό περίπου οι θέσεις ε, εργασίας ε, και οι εγκαταστάσεις και επίσης ε, πρέπει να πω ότι οι άλλες 130.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν από παρεμφερείς και παράπλευρες απώλειες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Θα πρέπει επίσης να δούμε την έννοια που αποδίδουμε στο μη ανταγωνιστικά ε, ορυχεία. Ε, δεν υπάρχει ο όρος αυτός σε κάποιο νομοθετικό κείμενο. Από το 2006 στο 2008, γιατί αυτές είναι οι τελευταίες μας ε, μετρήσεις, ε, δεν ε, είχαμε ακόμα μεγαλύτερο μέρος το, του άνθρακα από εισαγωγές παρά από την εγχώρια παραγωγή. Τώρα, το εάν υπάρχει συμβατότητα ανάμεσα στον άνθρακα και τις εναλλακτικέ μορφές ενέργειας, ε, ε, το ισπανικό παράδειγμα δείχνει ότι ναι, μπορεί να υπάρξει και ανάπτυξη του άνθρακα και ταυτόχρονη ανάπτυξη των ε, εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Το 2007 είχαμε 44.800 ε, ΜΒ ε, και κατά 18% ε, καλύφθηκε αυτό από άνθρακα, 16% από ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, έστω και αν το δυναμικό των ανανεώσιμων πυργών είναι τριπλάσιο από αυτό του άνθρακα. Αναφέρομαι στο 2008 που είχαμε το υψηλότερο ποσοστό αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια. Έχουμε επίσης προσαρμοστεί σε ένα άλλο ε, μείγμα, σε ένα άλλο είδος ε, άνθρακα που έχει λιγότερο οξύδιο του αζότου, έχει λιγότερο θείο κλπ. Ε, πρέπει να πω ότι έχουμε κάνει και ιδιαίτερες προσπάθειες έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν περαιτέρω μελέτες, έτσι ώστε να υπάρξει και περαιτέρω βελτίωση. Ε, στην Αστούρια, ε, όσον αφορά το θέμα στο οποίο αναφερθήκατε κύριε Καρβάλιο, ε, εμείς έχουμε το σύστημα της μετακαύσης. Είναι γεγονός ότι είναι πιλωτική η μονάδα. Έχουμε μια μονάδα 50 ΜΒ και θέλουμε να περάσουμε στα 300 ΜΒ στο μέλλον. Επίσης, σε σχέση με άλλα συστήματα, θεωρούμε ότι ε, αυτή η τεχνολογία είναι καλύτερη, γιατί μπορεί να προσαρμοστεί ε, σε ήδη φυστάμενες ε, μονάδες. Επίσης, τα κρατικά αποθέματα... Επίσης υπάρχουν χώροι για ενδεχόμενη αποθήκευση διοξιδίου. ε, αναφερθήκατε στην ιδιαίτερη κατάσταση της Ισπανίας όσον αφορά τον άνθρακα. Ε, εγώ μπορώ να σας πω ότι όλες οι αποφάσεις ε, της Ισπανικής κυβέρνησης είναι απολύτως συμβατές με την απόφαση 72-2007 του Συμβουλίου, τον κανονισμό συγγνώμη 72-2007 ε, του Συμβουλίου. Ε, έχουμε δώσει ένα χρονικό ορίζοντα του 2014 ε, για το κλείσιμο των μη ανταγωνιστικών ε, ορυχείων. Από την μία πλευρά συμφωνούμε με αυτό, από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να ακολουθήσουμε και τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέσπιση στρατηγικού αποθεματικού και επομένως δεν μπορούμε να οδηγούμε μόνο προς μία κατεύθυνση και όχι στην άλλη. Ευχαριστώ κύριο Πίκατς. E, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφερθώ σε ερωτήσει μία προς μία για την κυρία Καρβάλιο και τα σωματίδια. Ναι, είναι ένα τεχνικό ζήτημα, δύσκολο, όμως μια νέα οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές, τις οποίες υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ε, κάνει τους κανόνες εκπομπών πιο αυστηρούς. Με την τεχνολογία αυτή, ως αποτέλεσμα της αποθείωσης, θα μειωθούν οι εκπομπές σωματιδιών. Ο καθηγητής ο κύριος Γκέρεκ δεν είναι εδώ, αλλά δεν υπάρχει απαγόρευση οικοδόμησης ε, σταθμών ε, με άνθρακα με αποτελεσματικότητα πάνω από 50% απλά είναι πιο ακριβή αυτή τη στιγμή από τους άλλους. Τα υλικά που χρειάζονται για την κατασκευή τους είναι τόσο ακριβά ώστε δεν θα είναι ανταγωνιστική στην αγορά. Κατόπιν για το θέμα των ορυχείων. 117.000 άτομα απασχολούνται στην Πολωνία στα ορυχεία. Τα περισσότερα από αυτά είναι ανταγωνιστικά. Μιλάμε για τα 75 εκατομμύρια τόνους που εξορίχθηκαν είχαμε 100 εκατομμύρια επιδοτήσεις. Φέτος με αποτελεσματικότερες ε, μεθόδους εξόρυξης δεν θα χρειάζονται επιδοτήσεις καθώς θα είναι ανταγωνιστικά από μόνα τους τα ανθρακοριχεία. Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι, τόσα πολλά νοικοκυριά και οικογένειες που εξαρτώνται από την εξόριξη άνθρακα που δεν ε, μπορούμε να φανταστούμε πως η Πολωνία θα εγκαταλείψει την εξόριξη άνθρακα αυτή τη στιγμή και δεν χρειάζεται κιόλα. Όσον αφορά το κόστος ε, παραγωγής ε, ηλεκτρισμού με τη μέθοδο δέσμευση και αποθήκευση. Σύμφωνα με τους ειδικούς της εταιρείας μας, στην εμπορική φάση το κόστος δέσμευσης και αποθήκευσης θα είναι γύρω στα 35 ευρώ ανά τόνο δεσμευμένου διοξιδίου του άνθρακα. Εάν οι τιμές παραμείνουν όσο χαμηλές είναι αυτή τη στιγμή, η τεχνολογία αυτή δεν θα είναι ανταγωνιστική στην αγορά. Αλλά όταν μιλάμε για το κόστος δέσμευσης και αποθήκευσης, ξεχνάμε το πόσο επιδοτούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κάθε μεγαβατόρα ηλεκτρισμού από ΑΠΕ επιδοτείται με 30 και 40 ευρώ, στη δε Πολωνία με 70 ευρώ. Δεν βλέπω λοιπόν το πρόβλημα με το να επιδοτούμε τον ε, χαθαρό άνθρακα με 35 ευρώ. Γεγονό είναι πως είναι πολλά τα λεφτά δεδομένου του ποσοστού του άνθρακα στην παραγωγή ηλεκτρισμού αλλά ξεκολουθεί να είναι εφικτό. Γεγονός είναι πως οι τιμές σταδιακά θα ανέβουν και η δέσμευση και αποθήκευση θα γίνει πιο ανταγωνιστική. Προϋπόθεση είναι να περάσουν στην παραγωγή τα έργα επίδειξης για να βελτιωθεί η ε, τεχνολογία και να γίνει πιο φθηνή. Τέλος, Ακούστηκε το ερώτημα των Κρίστιαν Έλερ για το τι ελπίδα υπάρχει να εφαρμοστεί η οδηγία αυτή από τα κράτη-μέλη. Υπάρχει το ζήτημα της πολιτικής αποδοχής της ε, τεχνολογίας δεσμευσης και αποδοχής και διοικητικής αποδοχής. Δεν είναι γνωστή αυτή η τεχνολογία και υπάρχει ένα κλίμα φόβου και ανησυχούν ε, και είναι επιφυλακτική η πολιτική για την νέα αυτή τεχνολογία αλλά μόλις λειτουργήσουν τα έργα επίδειξης πρέπει να είναι έτοιμη η νομοθεσία. Αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συγχρηματοδοτήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις και τελευταίο σε αυτό το γύρο ο κύριος Γεξλέ. Και πάλι ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά ερωτήματα τέθηκαν, αλλά μέχρι το στιγμή δόθηκαν και πολλές απαντήσεις. Θα προσπαθήσω να προσφέρω επιπλέον απαντήσεις, αλλά αν παραλείψω κάτι το σημαντικό, επισημάνετε μου το στο τέλος. Πρώτον, ερώτηση για τα αποθέματα άνθρακα και για το ότι στη Νότια Αφρική έχουν μειωθεί, κάτι το οποίο δεν ανέφερα. Το νούμερο που ανέφερα είναι τα στοιχεία από την BGR, η γερμανική αρχή, που θεωρείται ενδεχομένως η καλύτερη πηγή τέτοιων στοιχείων. Επίσης, τέτοιο το θέμα για τον πόρων του άνθρακα ε, που υπάρχει ε, και είναι πολύ ε, μεγαλύτερος από το απόθεμα. Δηλαδή, απόθεμα σημαίνει τι μπορεί οικονομικά να ανακτηθεί. Και κατά καιρού υπάρχει ποσότητα άνθρακα που μπαίνει στο απόθεμα ή βγαίνει από το απόθεμα. Εξαρτάται από την ε, υπάρχουσα υποδομή. Τα νούμερα για τον άνθρακα ποικίλουν από αρχή σε αρχή και επίσης ανάλογα και με το τι ε, θεωρείται απόθεμα και τι θεωρείται πόρος. Η BGR μας δίνει 144 χρόνια, η, BP είναι 119 χρόνια, η διαφορά είναι μεγάλη, αλλά εν πάση περιπτώσει η ποσότητα είναι μεγάλη επίσης. Υπάρχει αρκετός άνθρακας και ήθελα αυτό να το επισημάνω. Αρκετές ερωτήσεις έγιναν για το θέμα της απασχόλησης ε, στον τομέα του άνθρακα, κυρίως στην Ισπανία. Από τότε που ξεκίνησα να εργάζομαι στον τομέα των ανθρακοριχείων στο Ηνωμένο Βασίλειο, χάθηκαν περίπου 235.000 θέσεις εργασία σε αυτόν τον κλάδο και παρεμένουν περίπου 5.000. Άρα, για να βρούμε πώς αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, η καλύτερη εμπειρία υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, το θέμα είναι να είναι αρκετά ισχυρή η οικονομία, ώστε να μπορέσουν αυτοί που απολύονται, που δεν έχουν δουλειά, να μπορέσουν να ξαναβρούν δουλειά και βεβαίως τίθεται το θέμα της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. Παρά τα αυτά, αφού χάθηκαν αυτές οι θέσεις εργασίας ε, από τα ορυχεία στι Ηνωμένης Βασίλειο με τη μείωση του αριθμού των ανθρακοριχείων, το Ηνωμένο Βασίλειο έγινε ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς άνθρακα πριν από 4-5 χρόνια ήταν ε, ο τέταρτος μεγαλύτερος εισαγωγέας άνθρακα, τώρα μας πέρασαν η Ινδία και η Κίνα. Όμως πρέπει να προσέξετε ότι δεν υπάρχει κανένα περιβαλλοντικό όφελος με τη μείωση της απασχόλησης στην εξόριξη ή την παραγωγή άνθρακα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μην ξεχνάμε ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα που έχουν σχέση με τον άνθρακα δεν αφορούν την εξόριξη ή την παραγωγή αλλά την καύση και το να μειωθούν τα ε, ορυχεία και να εισάγουμε άνθρακα από άλλες περιοχές του κόσμου δεν επηρεάζει αυτό περιβαλλοντικά την Ευρώπη. Τώρα, TST ανταγωνιστικό ορυχείο ανταγωνιστικό ορυχείο σε κάποιο, μέχρι κάποιο βαθμό καθορίζεται το, ε, από το είδος των αποθεμάτων και τη γεωλογική, γεωλογία του. Έχει σχέση με τις καθελογικές ε, επενδύσεις, με το βάθος και τα Κάποια ορυχεία αυτή τη στιγμή είναι πιο ανταγωνιστικά από ότι κάποια άλλα. Δυστυχώς πολλά από τα ευρωπαϊκά ανθρακοριχεία δεν αποδεικνύονται από ανταγωνιστικά, όχι λόγω ελλείψεως τεχνολογίας, αλλά του εξαιρετικά μεγάλου βάθους και των δύσκολων συνθήκων. Ετέθηκε το θέμα της ποιότητας του άνθρακα στην Ευρώπη. Υπάρχουν μεγάλες ποικιλίε διακιμάστη στην ποιότητα σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να πούμε ότι οι μονάδες παραγωγής ενέργειας μπορεί να σχεδιαστούν έτσι ώστε να και είναι περίπου οτιδήποτε. Μιλάμε για την εκπομπή κλασικών ρήπων στη λειτουργία, και μέχρι τη λειτουργία των Λεβίτων. Μπορεί κανείς να πει ότι κάποιο καύσιμο μπορεί να υποκατασταθεί από κάποιο άλλο. Εν πάση περιπτώσει, οποιαδήποτε μορφή άνθρακα που παράγεται στην Ευρώπη με τη σωστή τεχνολογία μπορεί να καεί. Τώρα, όσον αφορά το CCS ετέθη συγκεκριμένη ερώτηση του επιχειρηματικού μοντέλου για την δέσμευση. Ε, αυτό το απίδησε είδος, ήδη, ο κύριος Πίκατς. Θα ρωτήσω το ίδιο ίδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ποιο είναι το επιχειρηματικό μοντέλο για αυτές ή για την πυρηνική ενέργεια και ποιο είναι και το ETS, αυτό το εργαλείο ε, ανταλλαγής των εκπομπών από μόνο του δεν είναι επαρκή για να καθοδήγησει τις επενδύσεις προς ε, τεχνολογίες μηδενικής εκπομπής άνθρακα ή μήπως όχι. Και οι περισσότεροι θα συμφωνήσουν ότι το CCS η τεχνολογία αυτή παρότι αφορά μεγάλου, μεγάλης έκτασης προγράμματα μπορεί να συγκριθεί. Επίσης καταγορήσατε τον Μίστερ Τζόνστον ότι έδωσε ε, μια ενίσχυση στον ε, τομέα του άνθρακα. Παγκοσμίω δεν χρειάζεται βοήθεια η βιομηχανία άνθρακα. Το μέλλον της είναι πολύ εξασφαλισμένο εκτός Ευρώπης. Επανερχόμαστε λοιπόν στο ερώτημα που έθεσα εγώ αν θέλει δηλαδή η Ευρώπη να ε, ενταχθεί σε αυτή την πορεία ή αν θέλει να βγει. Ακόμα και αν μπορούσε να μην χρησιμοποιεί ε, άνθρακα η Ευρώπη, η χαμένη σε αυτή την περίπτωση θα ήταν εκτός από την, τον κλάδο, θα ήταν και η ευρωπαϊκή οικονομία επειδή θα ήταν πιο ακριβά τα μέτρα περιορισμού της βλάβης στο κλίμα. προσπάθησα να απαντήσω στις ερωτήσεις, αλλά αν υπάρχουν ερωτήσεις που άφησαν να σας παρακαλώ μου το επισημάνετε. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Φτάσαμε περίπου στο τέλος, εκτός αν έχουμε κάποια έκπληξη. Ε, δεν είναι ακριβώς έκπληξη, γιατί περιμέναμε το Γενικό Διευθυντή και θα ή, θέλαμε να του δώσουμε την ευκαιρία να πει δύο λόγια κάτι ε, για τον άνθρακα. Δεν μπορεί να μιλήσει για τα άλλα θέματα. Θα πάρει όμως τώρα το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω τις ε, ομιλίες όλων των παρισταμένων. Τις παρακολούθησαν οι συνάδελφοί μου. Θέλω να πω δύο λόγια από την, άποψη, από την άποψη της Ευρωπαϊκής ε, ενέργειας και σε σχέση και με την τεχνολογία CCS. Uh, Ένα τέταρτο της ηλεκτρικής μας ενέργειας προέρχεται από τον άνθρακα. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι πολλά κράτη-μέλη και θεωρούν τον Αθρακίτη και τον ε, Λιγνίτη ε, ως ε, σημαντικές πηγές εξασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασμού. Υπάρχει εσωτερικός, εσωτερική παραγωγή σε πολλά σημεία των κρατών μελών, ενώ έχουμε και εισαγωγές από διαφοροποιημένες αγορές τα αυτά, 80% των ε, εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προέρχονται από ε, την παραγωγή ενέργειας και βεβαίως ε, κυριαρχεί η παραγωγή διοξείδου του άνθρακα από την καύση του άνθρακα. Έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο μας δέσμευσε να μειώσουμε τα αέρια του θερμοκηπίου συνολικά στην οικονομία από το 85% στο 90% ε, με κάποια, μέχρι κάποια προθεσμία. Είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο είναι ουσιαστικό ουσιαστικά να αντιμετωπιστεί το θέμα της μείωσης των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου σε σχέση με τον άνθρακα. Είναι μεγάλη εμπειρία των παραγωγών άνθρακα σε καλές πρακτικές που μπορούν να μειώσουν την ένταση και να βελτιώσουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Όμως πολλά πρέπει να γίνουν. Κρίσιμη πρόκληση αφορά την, ε, τις τεχνολογίες CCS, οι οποίες καταρχήν ε, ήταν πολλά υποσχόμενες, αλλά βεβαίως η Ευρώπη πρέπει να δουλέψει για να υλοποιηθούν αυτές οι υποσχέσεις. Υπάρχει μια τεχνολογική δυσκολία, μια εμπορική δυσκολία και βεβαίως ε, το θέμα της αποδοχής τους από την ε, κοινή γνώμη και για την δέσμευση αλλά και την αποθήκευση του άνθρακα. Πρέπει και αυτά να τα κοιτάξουμε ε, προσεκτικά, να τα μελετήσουμε. Είναι σαφές ότι αν θέλαμε αυτές οι τεχνολογίες να συνολικά να πετύχουν, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να πετύχουμε τις ε, προγραμματισμένες μειώσεις. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά αφιέρωσε περίπου 15 ε, δις ευρώ στο σχέδιο ανάκαμψης για την ε, πρόθεση αυτών των τεχνολογιών και πρέπει να περιμένουμε και κάποια έσοδα από το ETS. Είναι σαφές ότι αυτό θα συνεχίσει να εντάσσεται στη στρατηγική του 2020 που θα προτείνει και θα εγκρίνει αύριο η Κομισιόν. Η στρατηγική θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας το Δεκέμβρη και προσβλέπουμε στην έκθεση του Κοινοβουλίου ε, στο ενδιάμεσο έγγραφο που συντάχθηκε ε, καθοδόν προς αυτή την ενεργειακή στρατηγική. Πρέπει εδώ να υπογραμμίσω ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική δεν προσεγγίζει την ενεργειακή πολιτική μελετώντας τα διαφορετικά κάψιμα και εντοπίζοντας τομέας προτεραιότητας ε, ε, εντόπισε τις προτεραιότητες όπως είναι η υποδοτικότητα της ενέργειας, προστασία των καταναλωτών, η, το να παραμείνουμε ε, ηγέτες σε κάποιους τεχνολογικούς τομείς και αναπτύσσοντας κάποια ε, ξεκάθαρη εξωτερική διάσταση στην πολιτική μας. Γιατί συμβαίνει αυτό, επειδή το ενεργειακό μείγμα κυρίως είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί σε εθνικό επίπεδο με την κοινή γνώμη ενώπιον των κοινοβουλίων με τις κυβερνήσεις και ακριβώς γι' αυτό η Κομισιόν ακολουθώντας αυτή τη στρατηγική θα ενημερωθεί πλήρως για τις συζητήσεις που γίνονται για το ενεργειακό μείγμα, πυρηνικό, άνθρακας με CCS, αέριο με CCS και ένα μεγάλο ποσοστό ανανεώσιμων. Και όλα αυτά θα ε, φανούν στον οδικό χάρτη εν του 2050 που θα παρουσιάσουμε το πρώτο εξάμεινο του 11. Αυτός ο δικός χάρτης δεν θα ε, προκύψει με βάση κάποια συνταγή τα διάφορα σενάρια πρέπει να μελετηθούν πιστεύουμε και από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο και να περιλάβουν ε, στο ενεργειακό μείγμα τις φιλοδοξίες και τις αποφάσεις που θα προκύψουν από τις εθνικές συζητήσεις που γίνονται τώρα και μόνο μέσω μιας πραγματικής ε, ε, πορείας, ε, προοδευτικής πορείας θα μπορέσουμε να πετύχουμε με τις πολιτικές μας. Αν με τις σωστές πολιτικές συμπεριλαμβανομένων και των προσπαθειών να βρούμε πηγές οικονομικά και ενεργειακά ε, αποδεκτές, θα μπορεί το CCS να παίξει σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό μείγμα. υπάρχουν και προϋποθέσεις, υπάρχουν δυσκολίες και βεβαίως ε, Υπάρχει και το τεχνολογικό εμπορικό σκέλος, το θέμα της αποδοχής από την κοινή γνώμη και ο βαθμός στον οποίο η εθνική προπολογισμού, όπως και σε άλλους τομείς νέων τεχνολογιών, ε, οι ανανεώσιμες κλπ, να στηρίξουν την στήριξη στον τομέα έρευνας ανάπτυξης αλλά και εξέλιξής τους. Είναι σαφές ότι ο στόχος της αφαίρεσης του άνθρακα θα απαιτήσει συνεχή προσπάθεια σε όλους τους τομείς, είτε ε, πρόκειται για CCS, τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια ή άλλε φιλικέ προ το περιβάλλον μορφέ ενέργεια. Αυτά έχω να πω, κύριε Πρόεδρε. Θα επανέλθουμε οπωσδήποτε στο ζήτημα αυτό ε, στι εκθέσει αναφορά ε, πρόοδου σχετικά με την κατάσταση της χρηματοδότησης των έργων αυτού του τομέα. Υπάρχουν κάποια έργα επίδειξης που αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούνται έξι αν δεν κάνω λάθος ε, τέτοιου είδους ε, έργα. Πράγμα που καταρχήν θα πρέπει να προσφέρει σωστή στήριξη στο στόχο να ε, αποκτήσουν εμπορικότητα γρήγορα. Αλλά βεβαίως αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες. Ευχαριστώ. Äh, ε, σας ευχαριστώ κύριε Λό, ευχαριστώ τους συναδέλφους, ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας, ευχαριστώ όσους μας έδωσαν ιδέες των Κριστιαν δηλαδή για αυτή την ακρόση. Καλό βράδυ, τέλος για σήμερα, ευχαριστώ.